Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας περάσουμε στην απογευματινή μας, λοιπόν, συνεδρίαση. Και αρχίζουμε με το σημείο 18. Ε, πρόκειται για μια διεξοδική ανάλυση του θεματικού τμήματος με θέμα τη σύμβαση για τις δικαστικές αποφάσεις. Μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή μας στα πλαίσια της διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Βασιζόμαστε στο σχέδιο σύμβασης του 2017 και θέλουμε να εξετάσουμε ποιες μπορεί να είναι επιπτώσεις στις διασυνοριακές διαφορές και την επίλυσή τους. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ μεταξύ μας τον καθηγητή Ασούνσιο, από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το Κομπουλτένσε, τον καθηγητή Κουνιβέρτη, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Για 20 λεπτά έχετε το λόγο και οι δύο μαζί, έτσι. Οπότε κανονίστε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω τη μελέτη αυτή ετοιμάστηκε από κοινού τον καθηγητή Κονιμπέρτη, εμένα και τον καθηγητή Σεν. Στην παρουσίασή μας θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη δομή. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθούμε στο πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της σύμβασης. Μετά θα ασχοληθούμε με την αλληλοεπίδραση της σύμβασης αυτής με άλλα διεθνή μέσα ε, τον κανονισμό των Βρυξελών 1 για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της σύμβασης σε διασυνοριακές διαφορές. Το σημείο κίνησης για μας είναι βασικό ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενοποίησει του κανόνε τη όσον αφορά την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, αλλά πρόκειται μόνο για αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων. Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες δηλαδή για δικαστικές αποφάσεις τρίτων χωρών. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας το πεδίο εφαρμογής, το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής στην αναγνώριση και την ε, θέση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Δεν πρόκειται για απευθεία κανόνες δικαιοδοσίας. Η αρχική ιδέα ήταν να καλυφθούν και οι δύο πτυχές, και η δικαιοδοσία δηλαδή και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, αλλά τελικά ε, καλύπτουμε μόνο το δεύτερο. Όσον αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογής, Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η σύμβαση εφαρμόζεται μόνο στην αμοιβαιότητα των αποφάσεων, δηλαδή μόνο στις αποφάσεις εκείνες με τις οποίες αποφασίζει να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμόζεται και στις χώρες που θα αποφασίσουν να προσχωρήσουν στη σύμβαση επίσης. Όσον αφορά το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογή, πρόκειται κυρίω για αστικά και εμπορικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσει, πώς είναι η νομική ικανότητα, διατροφή, οικογενειακά ζητήματα, κληρονομικά, αφαιρεγκαιότητα, μεταφορά αγαθών, ε, διαιτησία κλπ. Άρα το πεδίο εφαρμογής μοιάζει με εκείνο του κανονισμού ε, Βρυξέλλες 1, την αναδιατύπωσή του. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η δυσφήμιση εξαιρείται επίση, όπως επίσης υπάρχει δυνατότητα να εξαιρεθούν θέματα ιδιωτικού βίου και διανοητικής ε, ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα συνολικό πλαίσιο για την αναγνώριση και την ε, εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων τρίτων χωρών, θα υπάρχουν περιορισμοί από τη Σύμβαση. Πρώτα απ' όλα εξαιτία του περιορισμένου πεδίου εφαρμογή, αλλά επίση γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι αν δούμε τη σύμβαση της Χάγης, την προηγούμενη δηλαδή σύμβαση, λίγες πλευρές, η Σιγκαπούρη, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενταχθεί. Οπότε είναι άγνωστο πόσες χώρες θα συμφωνήσουν με τη νέα σύμβαση και θα προσχωρήσουν σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ε, αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων ε, τρίτων χωρών, ακόμα και αν είναι λίγες οι χώρες που θα συμμετέχουν και θα προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή. Εδώ έχουμε το περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης. Έχει να κάνει με την επιλογή των δικαστικών αποφάσεων και αναφέρεται και στην ε, μη αναγνώριση, την άρνηση αναγνώρισης και τις αιτίε που οδηγούν σε αυτήν. Κυρίως εδώ μας ενδιαφέρει το ότι η Σύμβαση προσπαθεί να δει ποια βάση δικαιοδοσίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή. Είναι επίσης σημαντικό εδώ να ξέρουμε ότι η Σύμβαση δεν ε, αποκλεί την εφαρμογή ενός μιας εθνικής διάταξης για την εφαρμογή εφόσον αυτή είναι πιο ευνοϊκή. Δηλαδή τα εθνικά συστήματα μπορεί να υπερισχύουν τη σύμβαση άπαξ και αυτή υπάρξει. Όσον αφορά τώρα τη σχέση με άλλα διεθνή εργαλεία. Εδώ έχουμε πολλές διεθνείς συμβάσεις που έχουν δημιουργηθεί αλλά είναι επίση αλήθεια ότι πολλά από τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν ε, με την προσπάθεια αποφυγής ε, αντίφασης με άλλες συμφωνίες. Υπάρχει αλληλεπίδραση πάντως με την επιλογή της σύμβασης του δικαστηρίου. Πρόκειται για μια ειδική σύμβαση που θα υπερισχύει. Η νέα σύμβαση δηλαδή δεν θα έχει άλλη επίδραση επί της προηγούμενης. Τώρα για να ταυτοποιηθούν θέματα διαφορών με άλλες συμβάσεις υπάρχει μια ευνοϊκή αναγνώριση των άλλων συμβάσεων, ακόμα και μελλοντικών. Υπάρχει ένα ευνοϊκό καθεστώς Υπάρχει μια ρήτρα μη επίδραση που θα είναι επίση πολύ σημαντική βάσει τη εφαρμογή τη σύμβαση του Λουτγκάνου και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει και ρήτρα αποσύνδεση. πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνει στους κανόνες ε, περιφερειακών ε, οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 α. Όσον αφορά τώρα την αλληλοεπίδραση με τον κανονισμό ακριβώς Βρυξέλλες 1, είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο του σχεδίου νέας σύμβασης δεν πρόκειται να υπονεμεύσει τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων του κανονισμού Βρυξέλλες 1 bis. δεν ε, θα είναι υποχρωμένη μια χώρα να δεχτεί αποφάσεις οι οποίες θα υπονομεύσουν ε, προηγούμενες ε, συμβάσεις. Και εξάλλου πολλές από τις διατάξεις είναι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στον κανονισμό Βρυξέλλες 1B με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με τους κανόνες που αφορούν τους καταναλωτές και τους υπαλλήλου, οι οποίοι προστατεύονται από αποφάσεις ξένων δικαστικών αρχών με υψηλό επίπεδο, όπως συμβαίνει και στον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Μπορεί να υπάρξει αναγνώρισή τους, αλλά συγχρόνως πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θα αποφεληθούν από τη δυνατότητα να μπορούν σε τρίτες συμβαλόμενες χώρες της μελλοντική σύμβασης αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του καταναλωτή. Στη μελέτη μας προτείνουμε κάποιες διευκρινήσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ανάλογα με το καθεστώς του Περιφερειακού Οικονομικού Οργανισμού μήπως μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες από τις διατάξεις σε χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής ε, Ολοκλήρωσης. Για τα υπόλοιπα, ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συναδέλφα και αγαπητέ πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή που προσθέναμε και πάλι στην Επιτροπή και θα συζητήσουμε το μοναδικό αντίκτυπο τη συνθήκη, τουλάχιστον του τι μπορούμε να προβλέψουμε στην παρούσα φάση για το μέλλον ε, της ε, θεματικής συνθήκης, της συνθήκης, συγγνώμη. Ε, σκοπός είναι να απελευθερωθεί η κυκλοφορία αλλοδαπών ε, δικαστικών αποφάσεων. Και άρα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της ε, συνθήκης είναι να δούμε κατά πόσο οι θα είναι πιο πιο φιλελεύθεροι ή λιγότερο φιλελεύθεροι σε σχέση με του μελλοντικού κανόνε που θα ισχύουν στα συμβαλαμένα μέρη. Αυτό θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καθορίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε του κανόνε που υφίστανται στη συνθήκη με του κανόνε που εφαρμόζονται στην παρούσα φάση από κάποια επιλεγμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη-μέλη. Και κράτη, συγγνώμη. Και φυσικά βασικό σκοπό είναι, σε την περίπτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση σε σχέση και με τι εξωτερικέ αποφάσει. Σημαντικό είναι να επιμείνουμε στο γεγονό ότι η πρακτική σημασία τη συνθήκη θα είναι ε, στο ύψιστο σημείο όπου χρειάζεται εφαρμογή από πρακτική άποψη. Αυτό ισχύει όταν μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν βρίσκονται στον τόπο όπου έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση. Για με άλλα λόγια, η δικαστική απόφαση του, της χώρας στην οποία ε, κατοικεί ο ενάγοντας δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η χώρα στην οποία θα έχει περιουσιακά στοιχεία ο ενάγοντας. Οι πιο σημαντικές λοιπόν αποφάσεις είναι αυτές που θα ληφθούν για δικοπραξίες που έχουν γίνει στο, στην Αλοδαπή και στη συνέχεια ο, το άτομο αυτό υπέτειος φεύγει από τη χώρα αυτή από την οποία έχει διαπράξει την αντικοπραξία, όπως για παράδειγμα η Facebook, η Google που είναι στην ε, Καλιφόρνια αλλά διαπράττουμε αντικοπραξία στην Ευρώπη ε, με έδρα όμω και περιουσιακά στοιχεία στην Καλιφόρνια. Θα πρέπει να εφαρμοστεί λοιπόν η δικαστική απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Καλιφόρνια. Και άλλη μία περίπτωση είναι η περίπτωση συμβάσεων που εκτελούνται στο εξωτερικό. Γι' αυτός λοιπόν τους, ε, σε αυτά λοιπόν τα δύο ζητήματα θα ήθελα να εστιαστώ. Ξεκινάμε λοιπόν στην προηγούμενη διαφάνεια για διάφορους λόγους με τις ΣΥΠΑ. Το δίκαιο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τις αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις είναι μάλλον συντηρητικό. Αυτό τι σημαίνει. Ότι είπα ΕΠΑ έχουν αυστηρές προδιαγραφές για να αναγνωρίσουν ε, αποφάσεις Χρειάζεται όχι μόνο να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του της αδικοπραξίας και της αλλοδαπής χώρας, αλλά και ο καθού να έχει πρώτερες δραστηριότητε στο κράτος μέλος αυτός. Είναι πιο δεσμευτικό και περιοριστικό αυτός κανόνας σε σχέση με το Βρυξέλλης 1 δις. Α. Και με τα όσα ισχύουν στα κράτη-μέλη είναι σημαντικό να επιμείνουμε λοιπόν σε αυτά, γιατί στην παρούσα φάση η συνθήκη αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα το δίκαιο των ΗΠΑ και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι βάσει αναγνωρίση άλλων δαπών δικαστικών αποφάσεων και τις ε, ο του Λεδαπού Δικαστηρίου ουσιαστικά ακολουθεί αυτές τις κριτικές ε, απόψεις που ισχύουν και στο δίκαιο των ΙΠΑ. Αυτό επίσης σημαίνει ότι από πολλές ε, πλευρές. Ε, η τρέχουσα συνθήκη για τους Αμερικανούς δεν είναι ούτε πιο φιλελεύθερη ούτε πιο συντηρητική σε σχέση με το Αμερικανικό δίκαιο. Είναι λίγο πολύ σε ίσο επίπεδο. Αντιθέτω, ε, το δίκαιο πολλών κρατών μελών, τουλάχιστον αυτά τα οποία εξετάσαμε και εμεί ε, στη μελέτη μα, πέντε στον αριθμό, είναι πολύ πιο φιλελεύθερο. Αυτό τι σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά το δίκαιο, για συνθήματα μάλλον δικαιοπραξιών και ε, κοιτάμε πού έχει διαπραχθεί ε, το, η αδικοπραξία, πού έχει προκληθεί η ζημιά από την αδικοπραξία που εκτελέστηκε στην Ελλαδάπη. Είναι λοιπόν πιο φιλελεύθερη η ζημια απο την αδικοπραξια που εκτελεστηκε στην ελλαδα ειναι λοιπον πιο φιλελευθερη η ερμηνεια των κρατών μελών. Και θα συνεχίσει να ισχύει αυτό, γιατί όπως είπε ο συνάδελφος, ε, πλέον στη συνθήκη υπάρχει μια πιο ευνοϊκή ρήτρα. Αυτό τι σημαίνει ότι ακόμα και αν ένα κράτος, ακόμα και αν συνθήκη είναι περιοριστική, τα συμβαλόμενα μέρη, τα κρατημέλη, θα εξακολουθήσουν να έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν ε, δικαστικές αποφάσεις σε περίπτωση πιο ευνοϊκού ε, εθνικού καθεστώτος. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι ότι μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση δεν πρόκειται να μετατροπεί αν εγκριθεί στην παρουσιαφάση ακόμα η συνθήκη οι ΙΠΑ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα και πολλά κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα πιο ευνοϊκά του καθεστώτα, ιδιαίτερω για δικαστικέ αποφάσει που προέρχονται για, από άλλε χώρε πέρα από τι ΗΠΑ. Αλλά το σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τι γίνεται σε άλλε χώρε. Υπάρχουν κράτη λοιπόν στον κόσμο τα οποία είναι πολύ πιο συντηρητικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ. Πιο συντηρητικά για διάφορου λόγου. Κάποια α, αρνούνται απόλυτα να εφαρμόσουν ε, αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις σε κάποιες χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία στην Ασία για παράδειγμα από ό,τι μου λένε. Κάποιες ε, ελέγχουν ε, και επαληθεύουν τις αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις όπως για παράδειγμα η Ινδία και ένας μεγάλος αριθμός κρατών μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία που ακολουθούν την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχονται μόνο δικαστικέ αποφάσει από χώρε ε, είτε στι οποίε ήταν παρόν να καθούν ε, κατά τη διάρκεια τη δικαστική απόφαση ή η οποία συνένεση στην δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου. Αλλά ερμηνεύουμε πολύ στενό τρόπο τι ρήτρε αυτέ. Είναι πάρα πολύ συντηρητικέ λοιπόν αυτέ οι χώρε και κάποιε είναι εντελώ κλειστέ σε ό,τι αφορά αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων. Είναι σαφέ λοιπόν ότι αν αυτά τα κράτη επικυρώσουν την το σχέδιο της συνθήκης, όπως έχει στην παρούσα φάση, θα ήταν πολύ σημαντική η βελτίωση για τα υπόλοιπα μέλη. Σημαντική λοιπόν η βελτίωση για τη ΣΥΠΑ, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα Αμερικανικά δικαστήρια θα ήταν ε, εφαρμόσιμα με πολύ πιο φιλελεύθερο καθεστώς στις χώρες αυτές που είναι κλειστές πλέον. Αυτό προφανώς είναι μια σαφής βελτίωση. Υπάρχουν και άλλα κράτη που έχουν μια προαπέτηση αμοιβαιότητας. Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι κυρίως στην Ασία, η Κίνα, η Ιαπωνία για παράδειγμα, αναγνωρίζουν μόνο τις αλλαταπές δικαστικές αποφάσεις στο βαθμό που η χώρα προέλευσης των αποφάσεων αναγνωρίζει και τις δικές τους ε, δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα λοιπόν με τις χώρες αυτές είναι ότι θα εφαρμόσουν τη συνθήκη μόνο και δεν θα χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πιο ευνοϊκών καθεστώτων σε σχέση με το εθνικό τους δίκαιο σε καλύτερο δηλαδή επίπεδο από ό,τι έχουμε στην παρούσα φάση από το σχέδιο της συνθήκης. Αυτό είναι κρίμα. Γιατί αν τα κράτη αυτά ήταν σε θέση και ήταν πρόθυμα να πάνε παραπέρα και να αποδεχθούν ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώ σε σχέση με αυτό που προβλέπεται στο σχέδιο τη συνθήκη, αυτό ενδεχομένω να ισχύει στην Κίνα, ξέρετε. Η Κίνα έχει συνάψει πάνω από 30 διμερεί συνθήκε με διάφορε χώρε σε όλο τον κόσμο και με κράτη, 9 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ τι διμερεί λοιπόν συνθήκε η Κίνα έχει αποδεχθεί τη βάση δικαιοδοσία πολύ πιο φιλελεύθερη από διατίθεται στην παρούσα φάση από το σχέδιο της συνθήκης της Χάγης. Άρα εδώ ενδεχομένως να υπάρχει περιθώριο για επιτεύξη συμφωνίας, ε, για μια πιο φιλόδοξη, πιο φιλελεύθερη συνθήκη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή, στην, στον κόσμο, όπως η Κίνα, ενδεχομένως όπως η Ιαπωνία και ορισμένες άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, και περνάμε στην τελευταία διαφάνεια, Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να διατηθούμε σήμερα είναι το εξή. Στην παρούσα φάση είναι σαφέ ότι η προτεραιότητα στι διαπραγματεύσει ήταν να αποκτήσουμε και να πετύχουμε τη συμφωνία των ΗΠΑ για να προσαρτηθούν, να προσαρτήσουν στην, στην ε, μελλοντική συνθήκη. Και αυτό εξηγεί γιατί η συνθήκη στην παρούσα φάση αποτυπώνει ουσιαστικά το Αμερικανικό δίκαιο. Είναι αυτό έχει δύο συνέπειες. Καταρχάς, το αποτέλεσμα είναι μία αρκετά χαμηλών τόνων συνθήκη. Με έλλειψη φιλοδοξίας. Δεν είναι τόσο σημαντική η πρακτική σημασία της. Γιατί δεν οδηγεί σε αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων από ένα δικαστήριο μόνο όταν έχει γυναική αντικοπραξία έχει υλοποιηθεί εκεί η σύμβαση ανεξάρτητα από τις ε, ε, δραστηριότητες του καθού. Εδώ θα χρειαζόταν να είχαμε την εφαρμογή αλλοδαπών αποφάσεων. Και στην παρούσα φάση η εφαρμογή των αλλοδαπών αποφάσεων δεν προβλέπεται από τη σύμβαση. Το δεύτερο θέμα είναι το εξή. Ενδεχομένω η ΕΙΠΑ τελικά να μην ε, επικυρώσουν την ε, σύμβαση. Είναι πολύ ενεργέ οι ΙΠΑ και στη Χάγη και εφαρμόζουν τι απόψει του, τι περνάνε με τα ζόρι, αλλά έχουν και ομοσπονδιακά ζητήματα στη ΣΥΠΑ που ενδεχομένω να οδηγήσουν τη ΣΥΠΑ να μην επικυρώσουν ποτέ τη σύμβαση αυτή ή αν την επικυρώσουν, να την επικυρώσουν σε επίπεδο πολιτιών. Οι πολιτείε δηλαδή να αποφασίσουν κατά πόσον θα την επικυρώσουν ή όχι. Άρα ένα σημαντικό ερώτημα είναι το εξή. Έχει νόημα να μπουν προτεραιότητε συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΑ και τελικά να υπάρξει έλλειψη φιλοδοξία στη σύμβαση και τελικά να έχουμε και μια σύμβαση που δεν θα την ε, επικυρώσουν οι ΕΠΑ. Υπάρχει μια εναλλακτική. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εναλλακτική, μια πιο φιλόδοξη σύμβαση ενδεχομένω μεταξύ ΕΠΑ και άλλων κρατών που θα, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διορθώνω, και άλλων χωρών που θα ήθελαν και αυτά πρόθυμα να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει διάφορα ασιατικά κράτη. Δεν θα συμπεριλάβει προφανώς τη ΣΥΠΑ. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η ΙΠΑ θα επικυρώσουν ποτέ τη σύμβαση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καθηγητή, για τα εισαγωγικά σας λόγια, και την παρουσίαση της ανάλυσής σας. Στρέφω προς τους ευρωβουλευτές. Θέλει κανένας να υποβάλει κάποιο ερώτημα, κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν τα κατάλαβα όλα σωστά. Κατά πόσον η συνθήκη της Χάγης στην παρούσα φάση ε, θα πρέπει να το θεωρήσουμε πιο πολύ, να τη θεωρήσουμε πιο πολύ ως πλαίσιο ένα πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται κάθε κρατός μέλος λίγο πολύ. Και δεν ξέρω κατά πόσον η σύσταση για διμερείς συνθήκες, για άμεση αναγνώριση και εκτέλεση ήταν αυτό που κατάλαβα σωστά. Ένα άλλο ερώτημα στο θέμα του Brexit. Σε τι βαθμό η Μεγάλη Βρετανία θα λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο την αναγνώριση και την εκτελεσιμότητα των αποφάσεων. Και εδώ ίσως να πρέπει να κοιτάξουμε την περίπτωση της Ιρλανδίας όλου του ιδιαίτερου. Υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώ ενδεχομένω να κινηθούν τα πράγματα. Αναφερθήκατε στην Google, στην προστασία των δεδομένων τα πράγματα έχουν ρυθμιστεί ως εξή. Χρειάζεται κάπως μία αντιπροσωπεία, ένα κατάστημα σαν ένα κράτος μέλος, προκειμένου για να μπορούμε να τους περιλάβουμε στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο αντιμετώπισης του θέματος στο μέλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι όποιο ασκεί εμπόριο της χώρας μας θα πρέπει να έχει μια κάποια αντιπροσωπεία η οποία θα είναι απόλυτα α, στην ε, δικαιοδοσία και θα ε, πρέπει να εκτελεί λοιπόν τις ε, αποφάσεις αυτές. Σε αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you very much. I do not have... Ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανένας άλλος το λόγο. Επομένως, οι δύο καθηγητές θα απαντήσουν τις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το αν η πρόταση είναι να εκπονηθούν διμερείς συμφωνίες ή όχι, με βάση την ανάλυση είναι ότι θα αξιολογήσουμε ε, την πρόταση σύμβασης και για να είναι επιτυχής η ολοκλήρωση της σύμβασης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η συνεισφορά της είναι πολύ περιορισμένη με την έννοια ότι λίγα κράτη συμμετέχουν στη σύμβαση. Και δεν θα μας εξασφαλίσει ένα γενικό σύστημα εκτέλεσης, αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων ε, γενικό, αλλά μόνο των κρατών που είναι συμβαλόμενα μέρη. Ε, και για τα κράτη τα συμμετέχοντα θα είναι δεσμευτικό εργαλείο, όπως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το περιεχόμενο ε, περιορίζεται και επηρεάζεται από την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να δούμε αν είναι λοιπόν δυνατόν να έχουμε μια πιο φιλόδοξη πρόταση, γιατί τα, οι κανόνες για την αρμοδιότητα ε, συμπεριλαμβάνουν κάποιες διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Δεν προβλέπεται επίσης η σύναψη διμερών ε, συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορες ε, εναλλακτικέ λύσεις. Ένα είναι να ρυθμίσουμε στην εσωτερική νομοθεσία μέσω κανονισμών ή κανονισμού την αναγνώριση των ε, αποφάσεων τρίτων χωρών και έχει αρμοδιότητα για να συνάπτει επίσης ε, διμερείς συμφωνίες και μην ξεχνάτε ότι η διάσκεψη τη χάγη είναι ένα πολυμερέ επίπεδο, πολυμερή σύμβαση. Μία πολυμερή σύμβαση έχει πάντα σημαντικούς περιορισμούς. Ε, λόγω ακριβώς του πολυμερούς χαρακτήρα της. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του Brexit, σε αυτή τη σύμβαση είναι σίγουρο ότι στο βαθμό που αυτή η σύμβαση ε, τελεσφορήσει και δώσει πραγματικά αποτελέσματα, γίνει μια πραγματική σύμβαση, τότε η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωριστά του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θα εξασφαλίσει ένα πλαίσιο για την εκτέλεση των αποφάσεων και θα υποκαταστήσουν μέρη ε, διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Για τη σύμβαση αυτή ε, πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ε, την σύμβαση του 2005 για την επιλογή του δικαστηρίου. Μιλάμε για αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Είναι περιορισμένη λοιπόν αυτή η σύμβαση του 2005. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και τη σχετική ερώτηση, η σύμβαση αποκλείει από το πεδίο εφαρμογή τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συκοφαντία και τα δικαιώματα στην ιδιωτική σφαίρα. αναφέρεται ρητά το privacy, ότι ε, εξαιρείται τα θέματα προστασίας των δεδομένων δεν είναι εντός της σύμβασης. Δεν είναι να αναγνωριστεί μία απόφαση τρίτης χώρας για να εκτελεστεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μηχανισμούς αμοιβαίας ε, εκτέλεσης. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω, να ρωτήσω. Όταν μιλάτε για την πιθανή προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση, σημαίνει ότι κατά την άποψή σας εδώ μιλάμε για τομέα αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Ναι, πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ε, ομιλητές, επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 19, που είναι μια δημόσια ακρόαση για, για το σχέδιο αποφάσεων της Χάγης. Ακούσαμε την παρουσίαση της μελέτης μόλις τώρα για τη διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές και τις αποφάσεις που εξετάζονται στα πλαίσια της διάσκεψης και τώρα θα περάσουμε στη σύμβαση, στην ακρόαση και θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες για το σχέδιο αποφάσεων της Χάγης. Καταρχάς, θα πάρουν το λόγο οι τρεις εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Just, της Κομισιόν, ε, η κυρία Ελβίνα Μορκίτε, ο κύριος Νόρελ Ρόσνερ και η κυρία Ανδρέα Σούλτς, αν προφέρω σωστά τα ονόματα. Για τις, θα, θα μας μιλήσω για τις διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμα, είναι εξελίξη. Έχετε 15 λεφτά όλοι μαζί. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Θα παρουσιάσουμε σύντομα το σχέδιο για τις αποφάσεις, θα μιλήσουμε για τις ε, ενεξελίξει διαπραγματεύσεις στη διάσκεψη της Χάγης, θα εστιάσουμε στα όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής και τι είναι ακόμα εκρεμές και ανοιχτό. Το σχέδιο για τις αποφάσεις, όπως ξέρουμε, είναι ένα σημαντικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγνώριση τη διαπραγματευόμαστε στη διάσκεψη της Χάγης επί τη βάση διαπραγματευτικών οδηγιών που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το 2016, όπως αναφέρθηκε ήδη στην προηγούμενη παρουσίαση, το σχέδιο για τις αποφάσεις ξεκίνησε το 1992 και οδήγησε στην υιοθέτηση τη Συμφωνία τη Χάγη του 2005 για την επιλογή του δικαστηρίου περιορισμένη πεδίου εφαρμογή. Επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 αυτή η σύμβαση. Και το 2012 το σχέδιο για τις αποφάσεις επανεκκινήθηκε. Ε, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας ε, που ολοκλήρωσε τις εργασίες για την ε, αναγνώση και εκτέλεση των αποφάσεων το τέλος του 2015 ε, και έχουμε το κείμενο λοιπόν του σχεδίου σύμβασης. Τα θετικά αποτελέσματα της ομάδας εργασίας επετέφθηκαν μετά από πέντε συνεδριάσεις. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάσκεψης της Χάγης το ε, συγκάλεσε μια ειδική επιτροπή για να ετοιμάσει ένα σχέδιο σύμβασης. Η ειδική επιτροπή λοιπόν συγκλήθηκε και για να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου. Συνεδρίσε τρεις φορές η Ειδική Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2016, τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2017 και τώρα θα συνεδριάσει το Μάιο του 2018 με σκοπό να οριστικοποιήσει το σχέδιο της σύμβασης και να υποβάλει το κείμενο αυτό στη διπλωματική διάσκεψη προς υιοθέτηση. Η διπλωματική διάσκεψη θα γίνει στα μέσα του 2019. Έχει ε, εγκριθεί το, το χρονοδιάγραμμα από το Συμβούλιο της Χάγης και στη διάσκεψη υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για αυτή την βασική νομοθετική προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από όλα τα μέλη της ε, διάσκεψης της Χάγης, λοιπόν. Η βασική στόχη της ε, σύμβασης αυτής είναι γενικά να ενισχύσει την ε, πρόσβαση πρακτικός πώς στη δικαιοσύνη μέσω της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αποφάσεων και να διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου, μειώνοντας το κόστος λόγω των ε, διασυνοριακών συναλλαγών. Όπως είπαν και οι καθηγητές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μια νομοθεσία αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων τρίτων χωρών. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει νομικές ε, αβεβαιότητες και να δικαίου και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει επιτυχής μηχανισμός για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων. Επομένως, ο πιο απλός τρόπος για να διορθώσουμε αυτή την έλλειψη νομικής ασφάλειας είναι να δουλέψουμε σε πολυμερές επίπεδο. Είναι το καταλληλότερο επίπεδο, πιο κατάλληλο από το ενωσιακό επίπεδο. Και είναι πιο αποτελεσματικό προφανώς από το διμερές επίπεδο. Το να δουλέψουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε σε πολυμερές επίπεδο να πετύχουμε κάτι τέτοιο, θα μα εξασφαλίσει παγκοσμίω τη δυνατότητα να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ευνοϊκό και για τους πολίτες αλλά και για τις εταιρείες της Ένωσης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά δικαστήρια με αυτόν τον τρόπο θα αναγνωρίζονται ε, από τις τρίτες χώρες ε, σε περίπτωση που είναι συμβαλόμενα μέρη. Αυτά είναι εισαγωγικά σχόλια και τώρα ο συνάδελφος θα συνεχίσει για τα επόμενα. Δηλαδή τι, έχει ήδη και τι έχουμε συμφωνήσει και τι μένει να γίνει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ πολύ που αναλάβατε την πρωτοβουλία να οργανώσετε την ακρόαση αυτή για αυτό το σημαντικό σχέδιο. Όπω είπε και η συνάδελφο, συνεχίζεται το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε δύο χρόνια που δουλεύουμε πάνω στο σχέδιο σύμβασης. Τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα. Η σύμβαση αυτή θα προσφέρει ένα σύνολο υποχρεώσεων για την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από άλλα συμβαλόμενα κράτη, αλλά και μια πιο ευνοϊκή ε, αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπό το εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει. Εξαιρούνται κάποια θέματα βέβαια. θα εφαρμόζεται σύμβαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με εμπορικέ συμβάσεις, ε, απασχόληση, αλλά με μεγάλη προστασία στο πιο αδύναμο μέρος, καταναλωτές, εργαζόμενοι, όταν μια εκτέλεση δικαστικής απόφασης είναι σε βάρος τους. Η σύμβαση έχει να κάνει με δικαστικές αποφάσεις, είτε διατάγματα είτε οτιδήποτε άλλο, καλύπτει και ε, διακανονισμούς δικαστικούς, αλλά όχι μέτρα προστασίας. Η σύμβαση συγχρόνως θα δημιουργήσει ένα σύστημα που θα προσφέρει αναγνώριση και εκτέλεση ξένων δικαστικών αποφάσεων εάν το δικαστήριο προέλευσης αποφάσισε βάση δικαιοδοσίας που αναφέρεται στη σύμβαση. Πρόκειται για την έμεση δικαιοδοσία. Το δικαστήριο πάντως, από το οποίο στείλει απόφαση και να την εκτελέσει, θα μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση και την εκτέλεση σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με τη δημόσια πολιτική ή με τις παραβιάσεις κάποιων διαδικαστικών κανόνων που έχουν να κάνουν με τον καθού, την ε, αποτυχία να προσφέρει ας πούμε το έγγραφο που αφορά τις διαδικασίες ή δεν έχει ο και το χρόνο στη διάθεσή του για να μπορέσει να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Συγχρόνως, η σύμβαση φροντίζει για την ευελιξία που μπορεί να χρειάζεται για να πετύχουμε ευρύτερη επικύρωση. Αποκλεί από το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα, μέσω δηλώσεων ειδικά θέματα όπου κάποια χώρα μέλος μπορεί να έχει ιδιαίτερο συμφέρον να μην εφαρμόσει την ε, σύμβαση στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται για θέματα που παραμένουν ακόμα σε κρεμότητα. Και θα δώσω το λόγο στον Ανδρέα Σούλς για τη συνέχεια. Στην Ανδρέα Ευχαριστώ πολύ και από μένα και καλησπέρα σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι στην ακρόαση αυτή, αυτό το σημαντικό πρόγραμμα. Δεν είναι η πρώτη ακρόαση που κάνετε γι' αυτό και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε και τελευταία η σημερινή όσο εξελίσσεται το κείμενο. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που παραμένουν σε κρεμότητα. Το πιο σημαντικό τεχνικά μιλώντας είναι το κατά πόσο οι διαφορές που έχουν να κάνουν με την διανοητική ιδιοκτησία θα συμπεριληφθούν ή όχι στο κείμενο της σύμβασης. Και παραμένει σε κρεμότητα γιατί διάφοροι ενδιαφερόμενοι για τη διανοητική ιδιοκτησία ενημερώθηκαν πολύ αργά για το πρόγραμμα αυτό και ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσει την ευκαιρία να σχηματίσουν άποψη. Συνεπώ προβλέπουμε σε έγγραφο το οποίο ετοιμάζει τώρα η διάσκεψη της Χάγης για ε, την νομοθεσία όσον αφορά την ε, διανοητική ιδιοκτησία για να δούμε στη συνέχεια πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα από την Σύμβαση. Υπάρχουν μόνο κάποιες προκαταρτικές απόψεις και αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μόνο τη δυνατότητα συμπερίληψης ή μη ε, στο τωρινό κείμενο για να διευκολύνουμε έτσι τις διαβολεύσεις. Γιατί αν δεν υπάρχει τίποτα στο κείμενο, οι διαβουλεύσεις θα ήταν πολύ δύσκολες. Πάντως θα υπάρξει, όπως είπαμε, το Μάιο συνεδρίαση της ειδική Επιτροπής και εκεί δεν θα συμπεριληφθεί αυτό το θέμα, δεν θα συζητηθεί. Και σίγουρα όχι διατάξεις που είναι σε παρένθεση τώρα. Γιατί θέλουμε να υπάρξει μια καλή και σωστή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ισχύει γενικότερα στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Όλες οι αντιπροσωπείες δηλαδή ένιωσαν ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να βρουν λύση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Πάντως, προς το παρόν οι απόψεις των διάφορων χωρών είναι διαφορετικές. Άλλοι θέλουν οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν οι διαφορές που έχουν να κάνουν με τη διανοητική διεκτήση και άλλες δεν το θέλουν καθόλου. Ελπίζουμε πάντως όσο προχωρήσει η συζήτηση να καταλήξουμε κάπου. Επίσης χρειάζονται περισσότερη συζήτηση για ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατά πόσο αποφάσεις δικαστηρίων που δεν είναι μιας μόνο χώρας, αλλά είναι κοινέ δικαστικές αρχές περισσότερων χωρών, πρέπει να αναγνωρίζονται υπό την έννοια της σύμβασης αυτής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για την διανοητική ιδιοκτησία όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει να κάνει και με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά ενδιαφέρει και άλλα δικαστήρια όπως είναι του Μπένελουξ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό. Για άλλε πάλι χώρε είναι ένα ζήτημα που του είναι εντελώ ξένο και άσχετο. Μια άλλη ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι η ρήτρα για τα μη ενωπημένα νομικά συστήματα. Δηλαδή πρόκειται για ομοσπονδιακές χώρες που έχουν διαφορετικές εδαφικές ε, οντότητες όπου σχήνουν διαφορετικές ε, διατάξεις. Αν κάποιος ε, κατοικεί δηλαδή σε μια χώρα, κατοικεί συγχρόνως και σε μια ενότητα της χώρας αυτής, οπότε τι ισχύει τότε δεν έχουμε αποφασίσει ούτε και κατά πόσο θα συμπεριλάβουμε το θέμα του κόστους των ε, διαδικασιών, της αναγνώρισης και της εκτέλεσης, για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Κυρίως όταν ε, κυκλοφορούν οι λεγόμενες cost orders, οι εντολές δηλαδή που αφορούν το κόστος των διαδικασιών αυτών. Για ορισμένους επίσης υπάρχει το θέμα του εμπορικού ή όχι που για ορισμένους πρέπει να αποκλείεται πλήρως, για άλλους όχι. Και αυτό πρέπει να λυθεί. Και όπως ακούσαμε και από τους δύο καθηγητές υπάρχει και το θέμα της συμπερίληψης ή όχι των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό βίο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζητάει γιατί το θέμα της δυσφήμισης εξαιρείται έτσι κι αλλιώς, αλλά η έννοια της δυσφήμισης ε, είναι διαφορετική σε διαφορετικά νομικά συστήματα. Υπάρχουν μερικά νομικά συστήματα που πιστεύουν ότι η δυσφήμιση είναι παραπληροφόρηση, ενώ για άλλους πρόκειται για σωστή πληροφόρηση. Οπότε η ερμηνεία είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί κάποιος να δώσει μια πληροφορία ε, χωρίς την άδεια του ενδιαφερόμενου και αυτό να θεωρηθεί δυσφήμιση για παράδειγμα. Και υπάρχουν και δύο ακόμα τεχνικά ζητήματα, αλλά πολύ σημαντικά. Τι θα γίνει αν ε, στα θέματα παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμα και αν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί τι κάνεις με το θέμα της εγκυρότητας ή όχι. Και εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο η διατύπωση προς το παρόν. Όλες οι αντιπροσωπείες φαίνεται να συμφωνούν ότι οι προηγούμενες συμβάσεις, οι πιο πρόσφατες, ε, μπορούν να περισχύουν τις σύμβάση και ο μόνος τρόπος, ή μάλλον το μόνο ζήτημα που μένει είναι πώς θα πετύχουμε στη διατύπωση να εκφράσουμε κάτι τέτοιο. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα συζητιόνται πάντως σε διάφορες άτυπες ομάδες εργασίας που το Μάιο θα ε, πούν τα βρήματα τους ποια είναι στην ε, Ειδική Επιτροπή. Πάντως αυτή η επόμενη Ειδική Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τη σύνταξη των διαφόρων ε, άρθρων που θα πάνε τελικά στη διπλωματική διάσκεψη και δεν θα ξανανοίξει το σχέδιο από την αρχή για όλα. Και θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο. Πέρα από το πρόγραμμα αυτό, και αυτό έχει να κάνει και με το πρόγραμμα εργασίας της διάσκεψης της Χάγης, γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και κάτι άλλο. Θέλουμε να εναρμονίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις ε, δικαιοδοσίες. Και συμφωνούμε για την αναγνώριση της πρώτης εκτέλεσης, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία, εφόσον υπάρξει συμφωνία πακέτου, ότι αργότερα θα γίνει μια προσπάθεια για την εναρμόνιση των κανόνων δικαιοδοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως κάναμε με το Βρυξέλλες 1α. Αυτά αποφασίστηκαν το Μάρτιο του 2016 και τα επανέλαβε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την ε, διάσκεψη της Χάγης φέτος. Πάντως φαινόταν ότι είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε και για τα δύο σχέδια συγχρόνως. Οπότε η ομάδα εμπειρογνωμόνων που κοιτάει την αναρμόνιση των κανόνων δικαιοδοσίας θα συνέλθει μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η, διπλωματική διάσκεψη για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων ξένων δικαστικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για τα μέσα του 2019. Ευχαριστώ, λέει και ο Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον, ε, στην κυρία Νίγκ του Ομοσπονδιακού Γραφείου της διάσκευή τη Χάγης. Ε, για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα ε, και ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας για το σημαντικό αυτό project. Πριν από δύο χρόνια ήταν εδώ ο συνάδελφός μου για να μιλήσει για το project αυτό το project δικαστικών αποφάσεων. Μετά από δύο χρόνια έχει προχωρήσει λοιπόν το έργο. Η σημερινή λοιπόν παρουσίαση βάσει και του ιστορικού υπόβαθρου που μας έδωσαν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα επικεντρωθώ λοιπόν σήμερα στο στόχο του project και στα ωφέλη του. να δώσω μια σύντομη εισαγωγή για την συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, την οργάνωση την οποία και εκπροσωπώ σήμερα. Έχετε κάποια ιδέα για την οργάνωση, φαντάζομαι. Μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος από το 2007. Η συνδιάσκεψη της Χάγης είναι μια διακυβερνητική οργάνωση. Από το 1893. Φέτος φορτάζουμε την 125η επέτειο. Έχουμε 83 μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη της συνδιάσκεψης της Χάγης και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρωτού περνάμε, περάσουμε στο project judgment να σας πω πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και την εκτελεσιμότητα γενικότερα. Γενικά, αντιμετωπίζεται στο εθνικό δίκαιο, σε αντιμερείς συνθήκε ή σε περιφερειακές και διεθνείς ε, διεθνικές συμφωνίες, όπως ο κανονισμός Βρυξέλλες 1. Άρα, Το θέμα που γίνεται για μια εταιρεία είναι τι γίνεται αν υπάρχει μια δικαστική επαφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται κατά πόσον ισχύει αυτό στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Καταρχά, η γενική απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ισχύουσα διεθνή ε, σύμβαση και εργαλείο. Άρα, η διάσκεψη της Χάγης θα είναι το κατάλληλο φόρουμ για την διαπραγμάτευση και τη συζήτηση των κοινών κανόνων Γιατί αυτή είναι η εντολή της διάσκεψης της Χάγης. Να προχωρήσει και να ενοποιήσει σταδιακά το εθνικό διεθνές δίκαιο. Οι καθηγητές μίλησαν για την ιστορία, το ιστορικό υπόβαθρο του project. Να σας πω ότι το 2005 είχαμε την επιλογή του δικαστηρίου της διάσκεψης. Εφαρμόζει μόνο αποφάσεις που έχουν λάβει τα μέλη η διάσκεψη. Έχουμε 80 μέλη λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μέξικο, Σιγκαπούρη και όλα τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης εξερμένης της ε, Δανίας Εκτός από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία που είναι, έχουν προσυπογράψει, να σας πω ότι η Κίνα και το Μαυροβούνιο προσυπέγραψαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και η Κίνα λοιπόν εργάζεται για να περάσει στην, υλοποίηση, στην ε, επικύρωση της ε, συνδιάσκεψης. Η Αυστραλία ε, επίσης και αυτή προετοιμάζεται για προσχώρηση. Και η Αυστρία. Η Αυστραλία λοιπόν ελπίζουμε να μπορέσει του χρόνου να προσχωρήσει. να επαναλάβω σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του project ότι το 2012 το Συμβούλιο της Συνήσκεψης Χάγης που είναι και το διευθυντικό όργανο έδωσε δύο εντολές. Η μία για μία ομάδα εργασίας για την αναγνώριση μάλλον για ένα project αναγνώρισης ε, των δικαστικών αποφάσεων και άλλη μία εντολή για τους κανόνες άμεσης δικαιοδοσίας. Θα σας πω αργότερα τι προέκυψε από τη συνάντηση των εμπρογνωμόνων. Μετά λοιπόν ε, από τις εντατικές εργασίες της ομάδας εργασίας, πλέον το project βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης και έχουν γίνει τρεις ειδικές συναντήσεις των επιτροπών. Η τελευταία, ελπίζουμε, θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου αν όλα πάνε καλά. Θα γίνει ένα σχέδιο από τη συνδιάσκεψη, το οποίο θα χορηγηθεί στους διπλωμάτες και τους περιογνώμονες. Θα επανέλθω σε αυτό στα επόμενα βήματα. Το project assessment είναι ένα βασικό project προτεραιότητας ε, δεν ξέρω βέβαια, μπορούν να προχωρήσουν οι διαφάνειες. Όχι. Αν θα μπορούσατε να προχωρήσετε, παρακαλώ. την επόμενη και την επόμενη διαφάνεια. στόχος λοιπόν της συνδιάσκεψης. Εγώ θα ήθελα να τονίσω απλά ότι βασικά είναι η προώθηση της ε, διεθνής ε, κινητικότητας μέσω καλύτερης ε, συνεργασίας με των εταιριών. Μεταξύ άλλων φυσικά και δικαστικής συνεργασίας για τη μείωση του κινδύνου σε περίπτωση προβλημάτων. σε σχέση με τη συνθήκη τη σύμβαση μάλλον του 2005. Είναι συμπληρωματική η συνδιάσκεψη. Αν και το 2005 ήταν ε, πολύ πιο ε, φιλόδοξη η συνδιάσκεψη. Και οι δύο λοιπόν αυτές οι συνθήκες προωθούν την αναγνώριση των αλληλοπών αποφάσεων. Η μελλοντική λοιπόν συνδιάσκεψη ε, θα έχει δύο βασικά ωφέλη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος του Σύμβαση και ένας πολίτης ε, λαμβάνει μια δικαστική αποφάση και αυτή είναι αναγνωρίσιμη σε άλλα κράτη-μέλη, αυτό τι σημαίνει ότι το άλλο μέλος θα χρειάζεται να ξεκινήσει δικαστικές ε, διαδικασίες και να κάνει αγωγή σε, άλλα, σε άλλες χώρες. Έτσι περιορίζεται το κόστος και περιορίζεται φυσικά και το χρονικό πλαίσιο. Άρα θα είναι πιο γρήγορη πρόσβαση στην δικαιοσύνη και πιο χαμηλή σε κόστος. Και θα βελτιωθεί και η προβλεψιμότητα του αποτελέσματος, μιας και ο Ευρωπαίος πολίτης θα είναι σε θέση να καθορίσει πιο σωστά τις συνθήκες για την αναγνώριση των αποφάσεων αυτό και να ξέρει με καλύτερο τρόπο πού θα ξεκινήσει να κάνει την αγωγή. Ένα άλλο όφελος θα αποτελέσει μια βασική συμβολή στο κράτος δικαίου και στο, στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους. Κάτι άλλο. Θα εξαχθούν, θεωρώ, οι δικαστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δικαστικές αποφάσεις του διεθνού ε, Εμπορικού Δικαστηρίου που έχουν ε, εκδοθεί από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Ολλανδικό, για παράδειγμα, σχετικό εμπορικό δικαστήριο. Αν συμπεριληφθούν λοιπόν αυτά και στη συνθήκη και τα θέματα διανοητική ε, περιουσίας, ε, τέτοιε ε, δικαστικέ αποφάσει θα περάσουν και τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί σημαντική συμβολή τη σύμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω επειδή θα υπάρχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, θα υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής των κρατών μελών για έντρα επίλυση των διαφορών στα επόμενα βήματα. Σύντομα θα έχουμε την ειδική αυτή επιτροπή, η οποία θα συζητήσει 7 βασικά θέματα προτεραιότητας τα οποία έχουν εντοπιστεί. Το θέμα της διανοητικής συντεκτησίας δεν θα συζητηθεί από την ειδική αυτή επιτροπή. Αν λοιπόν προκύψει ε, ένα σχέδιο σύμβαση από την ειδική αυτή επιτροπή, θα υπάρξει άλλη μια διπλωματική συνάντηση τον στα μέσα του 2019, η οποία και θα μας ε, επιτρέψει μετά από δύο-τρεις εβδομάδες να αναδιαπραγματευτούμε. Φυσικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευση όλων των ρητρών. Ελπίζουμε όμω να υπάρξει σύναψη τη συμφωνία τότε. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση τη ομάδα των εμπειρογνωμόνων για να εξετεθούν ζητήματα άμεση δικαιοδοσία. Όπω σα είπα, είχαμε δύο εντολέ το 2012. και η ομάδα των εμπειρογνωμών θα ξεκινήσει να κοιτάει τα θέματα τέτοια δικαιοδοσία. Κλείνοντα λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξή, ότι η διαδικασία, μάλλον το project judgment, θεωρώ ότι θα ωφελήσει ε, του Ευρωπαίου πολίτε και τι εταιρείε και είναι ένα στόχο τον οποίο αξίζει να πετύχουμε και σε ό,τι αφορά τα θέματα των ευρυστεχνιών σε θέματα τέτοια. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπέατρις Δεζέ. αν δεν απατώμε, με την προφορά του επωνύμου σας, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων. Παρακαλώ, έχετε 10 λεφτά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στους ε, Ευρωπαίους δικηγόρους. Να πω δύο λόγια, ε, προσωπώντας τους ε, δικηγόρους για αυτό το project επί του οποίου γενικά είμαστε θετικοί, ευνοϊκοί. Γιατί η αύξηση των ε, διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών ε, σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικότητα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εάν δεν έχουν ε, οι αποφάσει αν δεν είναι εκτελεστέ και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει εκτελεστότητα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το project μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση διεθνών διαφορών και μπορεί επίση να ενισχύσει την, τα κίνητρα για να προσφύγει κανείς ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Εάν τουλάχιστον ε, ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι αρμόδιο μέσω των δικαιοδοτικών φίλτρων που προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης. Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχουν παρόλα αυτά κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί μπορεί για τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών μπορεί να υπάρχει υποχρέωση να αναγνωρίσουν και να εκτελέσουν αποφάσεις οι οποίες προέρχονται από δικαστήρια τρίτων χωρών όπου οι δικαστικοί κανόνες και οι δικονομικοί κανόνες είναι λιγότερο υψηλοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτω ώστε οι λόγοι άρνησης να είναι επαρκώ ευρύ ούτω ώστε να μην αναγνωρίσουμε αποφάσει οι οποίε δεν έχουν εκδοθεί μέσα σε αποφάσει που είναι αντίστοιχε με τα δικά μα πρότυπα. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει γίνει πραγματικότητα, είναι στόχο. Ε, και για τον υπόλοιπο κόσμο είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Φυσικά δεν θα υπάρχει κοινή δικαιοδοσία για την ερμηνεία τη ε, σύμβαση, είναι πρόβλημα αυτό. Είδαμε τη σημασία που πήρε για την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, το θέμα της ερμηνείας των διατάξεων του καονισμού Βρυξέλλες 1, Βρυξέλλες 1α. Ε, μπορεί λοιπόν, κατά την άποψή μας, να δημιουργήσει αυτό, να αποτελέσει αυτό μια δυσκολία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγορικών ε, Συλλόγων γενικά θέλει μία προσέγγιση αρκετά ευρεία που θα αναγνωρίζει και θα εκτελεί τις αποφάσεις αλλά θα ε, συμπεριλαμβάνει και θέματα δικαιοδοσίας. Ε, υπάρχει όμως κίνδυνος να μην πετύχουμε κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε ότι ε, εν ώψη αυτού κινδύνου μπορούμε να περιοριστούμε στα θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τις εξαιρέσει για την έννοια της απόφασης. Συμφωνούμε με τον ορισμό. Φυσικά θα πρέπει να είναι σαφές ότι μια απόφαση δεν μπορεί να αφορά αποφάσεις ε, στις οποίες δεν εμφανίζεται ο καθού, δεν είναι παρόν. Είναι έμεσο, έμεσα αναφέρεται, έμεσα υπάρχει, αλλά καλό είναι να το διευκρινίσουμε στη σύμβαση. Το Συμβούλιο μας θεωρεί ότι καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν τα προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα, συντηρητικά μέτρα, εάν έχουμε ένα εξαρτητικό κατάλογο που τα προσδιορίζουν αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει φυσικά ο καθού να έχει δυνατότητα να εμφανιστεί φυσικός πώ και να έχει δυνατότητα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, εκκρεμοδικία, την ερημοδικία μάλλον, θα πρέπει να να σεβαστούμε την επίδοση του αρχικού κατηγορητήριου ε, της αρχικής αγωγής που υποβλήθηκε. Και βεβαίως ε, έχουμε και το άρθρο 7 με τους λόγους ε, άρνησης ε, που θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Επίσης, στα στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την εκτέλεση απόφαση υπάρχει η απόδειξη της επίδοσης της αρχικής αγωγής. Χωρίς αυτή την απόδειξη δεν υπάρχει αναγνώση και δεν υπάρχει εκτέλεση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει. Η δικαστικές ε, αποφάσεις ε, συμπεριλήφθηκαν υπό κάποιες προϋποθέσεις που απαριθμούνται σωστά στο σχέδιο σύμβασης. Στους αποκλεισμούς. Στις εξαιρέσεις. Ε, χαιρόμαστε για τη συμπερίληψη των ε, εργασιακών συμβάσεων και των καταναλωτικών συμβάσεων στο βαθμό που οι καταναλωτές και οι μισθωτοί έχουν κάποιες επιπλέον εγγύησεις σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη στη διαφορά, ε, τους υπόλοιπους διάδικους. Στο άρθρο 19 δηλαδή, του σχεδίου υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να βάλουν κάποιες ε, εξαιρέσεις σε περίπτωση σημαντικού εθνικού συμφέροντος. Νομίζουμε ότι το πεδίο εφαρμογής ε, που είναι πολύ περιορισμένο μπορεί μονομερός να, να περιοριστεί έτσι περαιτέρω από ένα συμβαλόμενο μέρος. Και έτσι θα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πεδίο εφαρμογής και δεν θα το θέλαμε φυσικά αυτό. Επίσης εγκρίνουμε την, ε, ε, τον αποκλεισμό της, διαδικασίας και όλων των, ε, της διατησίας και των διαδικασιών που αφορούν τη διατησία. Επίσης, η πιθανή εξαίρεση των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και ιδιωτική σφαίρα δείχνει τα όρια, τα σημαντικά όρια της σύμβασης και τους περιορισμούς της. Τώρα, για την αναγνώση και εκτέλεση των αποφάσεων, βλέπουμε ότι τα δικαιοδοτικά φίλτρα ε, βάζουν έμεσους κανόνες αρμοδιότητας. Μας αρέσει αυτό. Σε ό,τι αφορά τους ε, καταναλωτές και τους μισθωτούς, που είναι μέρη τα οποία θα πρέπει να προστατευθούν πολύ συγκεκριμένα αντί άλλων μερών, εναντί άλλων διαδίκων, σημειώνουμε ότι το δικαιοδοτικό φίλτρο προβλέπει ότι ο καθού θα πρέπει να, συνενεί με την αρμοδιότητα του αρχικού δικαστηρίου. Και αυτό θέλουμε εμείς να το αναφέρουμε ρητά, να αναφέρουμε ρητά δηλαδή ότι έχει ενημερωθεί ο καθού ε, και έχει δώσει την ε, συγκατάθεσή του πριν αναγνωριστεί και εκτελεστεί απόφαση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η ενοχικής υποχρέωσης. Η αναφορά στον τόπο όπου εκτελείται η υποχρέωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνεία, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 1α. Ο καθορισμός του τόπου εκτέλεσης της υποχρέωσης με βάση την συμφωνία των μερών θα πρέπει να τύχει απόφαση από τον, από τον δικαστή του προσώνει αίτηση κράτους. Μπορεί να δημιουργήσουν, ε, δημιουργηθούν ακαθόδη θέματα και να δημιουργηθούν συναφείς διαφορές. Επίσης για την εξαίρεση από αυτό το φίλτρο. Ε, όταν οι δραστηριότητες του καθού σε σχέση με την ε, συναλλαγή δεν είχαν καμία σχέση, τουλάχιστον εκ με το κράτος αυτό, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί η απόφαση να μην εκτελεστεί. τα δικαστήρια των συμβαλόμενων μερών μπορεί να κάνουν μια πολύ διαφορετική ερμηνεία. Ε, για το Συμβούλιο μας θα πρέπει να πλουστεύσουμε αυτές τις διατάξεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να πλουστεύσουμε αυτές τις διατάξεις. Μία από τις προτάσεις που κάνουμε είναι τουλάχιστον για την πώληση εμπορευμάτων και για τις ε, συμβάσεις υπηρεσιών που είναι οι ενοχές οι πιο σημαντικές και οι πιο συνήθεις στο παγκόσμιο εμπόριο, θα πρέπει να ξαναμπεί η διάταξη η οποία υπήρχε στο Βρυξέλλες 1α, για, ότι για την πώληση των αγαθών ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος ε, όπου παραδίδονται τα αγαθά ε, ή προσφέρεται υπηρεσίες πρέπει επίσης να, να αναφέρεται. Αυτές οι διατάξεις απλούστευσαν τον κανονισμό 1α και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλει αυτές οι διατάξεις να ενσωματωθούν τελικά στο σχέδιο της σύμβασης. Για τους λόγους αναγνώρισης και εκτέλεσης. Το Συμβούλιο είχε ζητήσει την συμπερίληψη άρνηση τη εκτέλεση. Είχε ε, ζητήσει την ε, συμπερίληψη των λόγων άρνηση που υπήρχε στη Σύμβαση Χάγηση ε, στι συμφωνίε για την εκλογή του δικαστηρίου. Βλέπουμε ότι κάποια αυτά τα κριτήρια έχουν συμπεριληφθεί, έχουν παραμείνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία παρατήρηση, είναι ότι στο αρθρο 7.1.D, με βάση το οποίο η αναγνώριση, η εκτέλεση μπορεί να μην γίνει, εάν η διαδικασία ενώπιον του αρχικού δικαστηρίου ήταν αντίθετη με, μη, με τόσο προβλέπει η συμφωνία ε, και επομένως η διαφορά έπρεπε να, να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο, θα θέλαμε να προσθέσουμε σε αυτή τη ρήτρα μία αναφορά που θα λέει εκτός και αν η συμφωνία ε, δεν υπάρχει με βάση ε, το δίκαιο του δικαστηρίου που έχει εκλεγεί με βάση το άρθρο 9 της Σύμβασης για τις ε, συμφωνίες ε, εκλογής δικαστηρίου. Άλλη παρατήρηση του Συμβουλίου μας είναι ότι οι λόγοι άρνησης ε, δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα το θέμα είναι λοιπόν μήπως θα πρέπει να τις κάνουμε, να τις καταστήσουμε αυτές, αυτούς τους λόγους μάλλον τους καταστήσουμε υποχρεωτικούς. Τελευταίο σημείο είναι ότι εγκρίνουμε τους λόγους άρνησης σε περίπτωση που η αποζημίωση και, τα, και η τόκοι είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Πάμε στην τελευταία διαφάνεια. Γενικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είμαστε είναι υπέρ του σχεδίου αυτού, αυτή τη σύμβαση, αλλά ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα υπεράσπισης και στα δικαιώματα ε, Επίση, Επίσης, ε, ο σεβασμός των ε, δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Πολιτών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια διαδικασιών που γίνονται σε τρίτες χώρες, ειδικά ε, να προσέξουμε το θέμα της, ε, ε, των ισότιμων δικαιοδοτικών κανόνων. Ε, αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος. Καλό τον, κυρία, τον κύριο Ηλία Κοντέα από την Business Europe που θα μας μιλήσει για την άποψη της δικιάς του οργάνωσης. Πρόκειται για την διανοητική ιδιοκτησία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου αποστήλατε. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο παθήθηκε ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή όχι στο σχέδιο αυτό σύμβασης. Όπως είπε και η Επιτροπή, ενημερωθήκαμε για τις συζητήσεις αυτές μόνο πέρυσι. Οπότε, ο αντίκτυπος μια τέτοια συμπερίληψης μας απασχόλησε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τώρα. Θέλω εδώ να αποσαφενήσω ότι εμείς δεν ζητάμε ρητά να συμπεριληφθεί η διανοητική ιδιοκτησία στο πεδίο εφαρμογή τη σύμβαση αυτή, γιατί δεν νιώσαμε ότι υπήρχε τέτοια ανάγκη. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι το σχέδιο αυτό έχει ένα μεγάλο στόχο, όμως σήμερα είμαστε κατά του να συμπεριληφθούν, αν μη τι άλλο, τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, τα σήματα και τα σχέδια στο πεδίο εφαρμογή τη σύμβαση. Είναι πολύ περίπλοκη η νομοθεσία για την δυνητική ιδιοκτησία, γι' αυτό φοβόμαστε ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με απρόβλεπε συνέπειε εφόσον συμπεριληφθεί. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, υπάρχει θέμα ερμηνεία διότι δεν υπάρχει δικαστήριο που να έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την ερμηνεία της Σύμβασης της Χάγης. Μέχρι τώρα, για να έρθω σε κάτι πιο συγκεκριμένο, ε, ποιο θα ήταν το πρόβλημα σε σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες και ποιες είναι αυτές την εκείνη των Παρισίων για την βιομηχανική διοκτησία που βασίζεται σε δύο βασικές αρχές. Το ένα είναι η επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο και το δεύτερο είναι η ανεξαρτησία των διπλωμάτων αεροσυντεχνία. Το πρώτο σημαίνει ότι κάθε χώρα μέλο ε, προσφέρει την ίδια προστασία και στους υπηκόους άλλων χωρών, όπως προσφέρει και στους ίδιους τους υπηκόους της, αλλά και τις ε, νομικές ε, διορθώσεις που απορρέουν από μια τέτοια συμπεριφορά. Υπό το σχέδιο όμως σύμβασης όσο έχει τώρα, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση των Παρισίων θα μπορούσε να υποχρεωθεί να εκτελέσει μια ξένη δικαστική απόφαση που σύμφωνα με το δικό της δίκαιο δεν είχε την υποχρέωση να εκτελέσει ή να εκτελέσει διαφορετικά. Έπειτα στο δεύτερο, που είναι η ανεξαρτησία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Αυτό αντικατοπτρίζει ακριβώ την εδαφική φύση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και επί ουσία σημαίνει ότι η τύχη ενό διπλώματο ευρεσιτεχνία σε μια χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την τύχη του ίδιου διπλώματο ευρεσιτεχνία σε κάποια άλλη χώρα. Έτσι όπω ε, αναφέρει σήμερα το σχέδιο σύμβαση θα, θα υπάρχει κανένα περιορισμός. Η ερμηνεία θα γίνεται χωρίς περιορισμό. Άρα η εκτέλεση μιας ξένης απόφασης σημαίνει αν μη τι άλλο να υπάρχει ρητή επιβεβαίωση ότι η, το λόγο δίπλωμα ευρεσιτεχνία έχει εγκριθεί με εγκυρότητα. Τώρα όμως υπάρχει η περίπτωση να περιοριστεί η ανεξαρτησία τη χώρα ε, εκτέλεση. Ιδιαίτερα ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση βρίσκεται σε εκκρεμότητα στη χώρα εκτέλεσης. Η χώρα εκτέλεσης έχει αρνηθεί να εφαρμόσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση, να έχει ανακαλέσει το δίπλωμα αυτό. Αργότερα, μετά τη Σύμβαση των Παρισίων, Είχαμε και άλλες συμφωνίες που υποχρένουν τις ε, συμβαλόμενες χώρες να εφαρμόσουν αυτή την αρχή. Οπότε τίθεται πάλι το ίδιο ζήτημα όπως έγινε με τα TRIPS. Κατά τη γνώμη μας, αν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ε, προσφέρει ελάχιστα ωφέλη. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορών για την διανοητική ιδιοκτησία, η λύση που θέλει συνήθως ε, ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων είναι η διαταγή πληρωμής. Υπάρχουν διαφορές στο ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο που έχει σαν αποτέλεσμα η αναγνώριση των διαταγών αυτών να μην είναι επιθυμητή. Γιατί ένα τέτοιο διακανονισμό θα ήταν επιθυμητό μόνο εφόσον υπήρξε ένα πλήρε αναρμονισμένο σώμα ουσιαστικού δικαίου με ευθυγραμμισμένε δικαστικέ διαδικασίε, που από ό,τι ακούσαμε μπορεί να γίνει, αλλά σε μετέπειτα στάδιο. Και είναι αλήθεια ότι μόνο σε ένα ενωπημένο τέτοιο σώμα μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και σε βαθμό που να ικανοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι ιδιοκτήτε δηλαδή οι διανοητική ιδιοκτησία. Προ το παρόν όμω δεν έχει δοκιμαστεί κάτι τέτοιο. Και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε κατά πόσο θα γίνει ποτέ πραγματικότητα μια τέτοια ενωπημένη διαδικασία έγκριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Οπότε όσον αφορά τα υφέλη, τα υφέλη, μόνο μια οικονομική αποζημίωση θα μπορούσε να εκτελεστεί. Οι περισσότερες περιπτώσεις όμως διανοητικής διαδικασίας ολοκληρώνονται πριν αποδοθεί αποζημίωση, εκτελεστεί. Άπαξ και το θέμα της διαταγής έχει αποφασιστεί με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θέματα που έχουν να κάνουν με αποζημιώσεις εκπίπτουν ή τέλο πάντων τακτοποιούνται. Δηλαδή το «φέλη» θέλω να πω φαίνεται ότι θα είναι πολύ περιορισμένα. Και μιλώντας με τα μέλη μας, δεν έχουμε υπόψη μας καμία περίπτωση όπου χρειάστηκε ε, ένας ε, ενάγωνο να φτάσει σε μια περίπτωση διασυνοριακά να εισπράξει τέτοια αποζημίωση. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα μηνύματα όσον αφορά σοβαρούς κινδύνους και επιδείνωση της κατάστασης. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα επίλυσης και μπορεί να υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την ερμηνεία και δεν θα υπάρχει τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ερμηνείας. Επίσης, αν υπάρξει περισσότερη, περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχουν εγγύησεις για τα ωφέλα. Συνολικά δηλαδή πιστεύουμε ότι θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη βεβαιότητα, ε, μεγαλύτερο κόστος για όλες τις επιχειρήσεις παντός ε, μεγέθους που θα εμπλακούν σε μια τέτοια περίπτωση διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι συζητήσεις βέβαια συνεχίζονται και εμείς προσβλέπουμε στη συνέχιση των συζητήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε ότι αναμένουμε ένα έγγραφο από τη Γραμματεία για τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οπότε αναμένουμε τα έγγραφα αυτά και να τα συζητήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση που να αντικατοπτρίζει και τις θέσεις των ενδιαφερομένων πλευρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα έχει έρθει η ώρα για ερωταπαντήσεις. Ο κύριος Φως. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και του προσκεκλημένου μα για τι παρεμβάσει του. Έχω διάφορε ερωτήσει να κάνω. Δεν σα υπόσχομαι ότι θα τι παρουσιάσω σε διαρθρωμένο τρόπο. Αλλά όποιο θέλει, απαντήσει. Άκουσα τα βασικά στοιχεία που με απασχολούν επί ποιων προτύπων θα πρέπει να στηρίξουμε την όλη διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Να ξεκινήσουμε με κάποια παρόμοια πρότυπα κατά νου, για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και το ερώτημα του πώς ε, θα υπάρξει μια κοινή ερμηνεία όλων των κανόνων αυτών. Και τι θα γίνει αν ένα κράτος δεν τηρήσει καν αυτές τις κοινέ ε, συμφωνίες. Θα υπάρξουν ε, κυρώσεις, θα υπάρξουν κριτήρια αποκλεισμού. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε υπόψη μας. Για την εκπρόσωπο της CCBA να ρωτήσω γιατί δεν θα πρέπει να παίξουν ρόλο τα διευθυντικά δικαστήρια. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, καθαρά για χρονικούς ε, λόγους, μπορούν να παίξουν ρόλο. Ή για να αποφύγουν παρανοήσεις σε άλλα επίπεδα. Και άλλες τρεις αν μου επιτρέπετε. Τι γίνεται με τις συλλογικές αγωγές Υπάρχουν και εδώ κάποιες ειδικές προδιαγραφές, κάποιες ιδέες, ενδεχομένως να υπάρχουν κοινά πρότυπα. Ή όταν ε, λαμβάνουν αποφάσεις να μπορούν να επεκτείνονται. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου οι πολιτισμικοί κύκλοι απομονώνονται και πάνε. Και εδώ τίθεται πάλι το θέμα των προτύπων και τι μπορούμε να κάνουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά κυρίω στον τομέα της, ε, του αστικού δικαίου έχουμε τρόπους ζωή σε άλλες πολιτισμικούς κύκλους που δεν μπορούν να τύχουν αναγνώριση σε μας ε, χωρίς ε, κάποια προσαρμογή, γιατί αποκλίνουν υπερβολικά. Ιδιαίτερα κοιτώντα τον τομέα του Ισλάμ. Εδώ υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε εντελώς ε, διαφορετικές βάσεις, σε πιο πολύ θρησκευτική φύσεως, που δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία των δικαστηριών και βρισκόμαστε και σε μια χρονική συγκυρία όπου αποφάσεις, οι αποφάσεις μπορούν να τύχουν κατάχρησης από κράτη-μέλη και να είναι πολιτικά τα κίνητρα πίσω από κάποια απόφαση. Έχω υπόψη μου για παράδειγμα στην παρούσα φάση στην Τουρκία, όπου όχι μόνο κατηγορείται κανεί για τρομοκρατία κατευθείαν μετά που θα βγει κάτι κατά του κράτου και τη κυβέρνηση, αλλά και Υπάρχουν λοιπόν ε, αντίπεινα και τελικά η δικαστική απόφαση καταλήγει να έχει πολιτικό υπόβαθρο. Με τα δικά πρότυπα λοιπόν αυτά δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορείτε να τα απαντήσετε όλα αυτά, αλλά αυτά με απασχολούν. σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά αυτά νομικά συστήματα με μια κοινή βάση και η εκτελεσιμότητα αυτών. θα πρέπει να δούμε ότι είναι πολλές οι πολιτικές ιδιαιτερότητες και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των διαφορών κοινωνιών και σε ό,τι αφορά τις συλλογικέ αγωγές θα πρέπει να δούμε τι ισχύει και τι μπορεί να ισχύσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ Όσου πήραν το λόγο εδώ, γιατί μας παρουσίασαν μια πλήρη εικόνα της κατάσταση πρόοδου όσον αφορά την διάσκεψη της Χάγης για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι προχωράμε προς μια κατεύθυνση κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων. πρώτη μου ερώτηση, αν καταλήξει κάπου αυτό. Θα μπορούσαμε όντω να μιλήσουμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων. Δεύτερον, κατάλαβα ότι είναι μια αρχή που χρειάζεται εξαιρέσεις. Με αιτιολογικά βέβαια. Έχουμε ήδη καταλήξει σε κάποιες λύσεις ή όχι για αυτές τις αιτιολογήσεις, έτσι, των εξαιρέσεων. Γιατί μπορεί να μας αρέσει οι αποφάσεις οι δικές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγονται στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά το αντίστροφο μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστικό. Και εκφράστηκε αυτή η ανησυχία από κάποιον. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει εξαίρεση, θα πρέπει η αιτιολόγηση να είναι αρκετά ισχυρή για να μην εφαρμόζουμε τέτοιες αποφάσεις. Έπειτα υπάρχει και το τιμωρητικό που φυσικά και δεν πρέπει να δεχτούμε. Και υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα που επίση έδωσε ο κύριος Φως. Υπάρχουν κάποιες θρησκευτικέ αρχές που μπορεί να επηρεάζουν το δίκαιο ορισμένων χωρών. Στις δικές μας χώρες δεν ισχύει αυτό. Οπότε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αυτή η αιτιολόγηση των ε, αρνήσεων εκτέλεσης με ενδιαφέρει. Και έρχομαι στην τρίτη μου ερώτηση. Εάν αυτή η αιτιολόγηση άρνησης οδηγήσει στο να περιθωριοποιούνται όντω οι αποφάσεις κάποιων αρχών, αυτό δεν θα υπονομεύσει τελικά την σύμβαση, γιατί δεν θα υπάρχει η αμεβαιότητα. Υπάρχουν οι μουσουλμανικές χώρες, εντάξει, αν κάθε φορά αρνούμαστε με την αιτιολόγηση που θα δίνουμε να εφαρμόζουμε τις δικές τους αποφάσεις, θα αρχίσουν και αυτοί να μην εκτελούν τις δικές μας. Κάποιος είπε ότι η Δανία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, οπότε ρωτάω, καλά το κατάλαβα, γιατί αποκλείεται η Δανία το έχει ζητήσει και γιατί, αν η απάντηση είναι ναι. Και τέλος, το πιο βασικό, η σύμβαση αυτή θα εφαρμοστεί εύκολα. Έχω κάποια αμφιβολία, γιατί δεν προβλέπεται κανένας μηχανισμός που να πιέσει τις εθνικές δικαιοδοσίες να ερμηνεύουν ομοιόμορφα τις αποφάσεις. Οπότε θέλει πολλή δουλειά από τις χώρες μέλη. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος οι ερμηνείες να είναι πολύ διαφορετικές. Πώς θα αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Και αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις. Προφανώς ε, δεν καλείστε να απαντήσετε σε όλες εξ αυτών. Επιλέξτε αυτές που σας ταιριάζουν πιο πολύ. Να απαντήσω έτσι συντομία στα ερωτήματα τα οποία τέθησαν προς τους δικηγόρους. Στα ρώτησε ο κύριος Φως. Πώς θα διασφαλίσουμε μια κοινή ερμηνεία, αν όχι ομοιόμορφη και άλλοι μπορούν να απαντήσουν εκτό από μένα βέβαια. Πάντω αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ε, το κάθε συμβαλόμενο μέρο μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο τις αποφάσει, αλλά υπάρχει μια νομολογία που δημιουργείται σιγά σιγά. Αυτό το έχουμε δει και με άλλε συμβάσει. Δυστυχώ, δεν είμαστε εξοπλισμένοι ώστε να πιέσουμε μια χώρα να εφαρμόσει μια απόφαση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη από τη δικιά μου, εντάξει. Τώρα για τη διαιτησία. Ήδη υπάρχει μια διεθνή σύμβαση που έχει να κάνει με τη διαιτησία και ήθιστε να αποκλείεται από αυτού του είδους εργαλεία, ακριβώς για να μην παρεμβαίνει. Τρίτο. Για να απαντήσω όσον αφορά την αιτιολόγηση άρνησης εκτέλεσης. Αν εφαρμοστεί ευρέως η σύμβαση αυτή, προφανώς θα εφαρμόζεται σε χώρες που έχουν και διαφορετικές παραδόσεις και συνήθειες. Στο σχέδιο σύμβασης υπάρχει πάντα η αιτιολόγηση διατήρηση δημόσιας τάξης, για παράδειγμα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 1α πρόκειται για πραγματικά εξαίρεση. Ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται ποτέ η εξαίρεση, είναι πολύ σπάνιο. Όμως στα πλαίσια αυτής της σύμβασης, κατά πάσα πιθανότητα, θα παραμείνει αιτιολογία άρνησης που θα χρησιμοποιείται πιο συχνά. Αν μου επιτρέπετε, να συνεχίσω εγώ τώρα. Για την ερώτηση του κυρία Φώσα. Ε, γιατί εξαιρείται η χώρα αυτή. Η συνθήκη της Νέα Υόρκης για την ε, εκτέλεση των ε, αποφάσεων των δικαστικών, των δικαστηρίων δεν θέλουμε να διακυβευθεί και έχουμε και τη σχετική ρήτρα στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 με πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογή. Ε, αυτό τι σημαίνει ότι οι αποφάσεις οι δικαστικές που υποστηρίζουν ένα δυτικό δικαστήριο και που αποσκοπούν, για παράδειγμα, στο διορισμό ενό ε, δυτικού δικαστή ή άλλα τέτοια προστατευτικά μέτρα, θα πρέπει να αποκλείονται, γιατί αυτό συγκαταλέγεται σε άλλο πλαίσιο και δεν θέλουμε να τα βάλουμε στην συνδιάσκεψη για το κατά πόσο υπάρχουν κυρώσεις, για το κατα... αν, μια χώρα δεν τηρήσει τους κανόνες ε, εκτελεσιμότητας. Ε, κυρώσει υπό την αυστηρή έννοια δεν υπάρχουν, αλλά η συνδιάσκεψη τη ΧΑΚΙΣ από το 1893 κάνει διεθνεί ε, συμβάσει. και ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται είναι ο εξής. Κάθε σύμβαση συνοδεύεται από μια επεξηγηματική έκθεση η οποία είναι παρόμοια με τα γερμανικά σχόλια σε, στα νομοσχέδια, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στη δικαστικό σώμα για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Και σε μία περίπτωση, α, μάλλον στην αρχή αναφέρεται η πρόθεση του νομοθέτη. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Έχουμε έναν εκπρόσωπο από το αστικό δίκαιο και έναν ε, εκπρόσωπο από το common law και κυρίως οι εκθέσεις αυτές ε, ψηφίσονται από τα κράτη. Δηλαδή, αν το κείμενο πρέπει να ερμηνευτεί, η ερμηνεία συγκαταλέγεται στο κείμενο. Για το κατά πόσον ε, πρόκειται για ελεύθερη κυκλοφορία δικαστικών αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα πως ναι. Αλλά δεν το έχουμε πετύχει αυτό ακόμα. Αλλά σίγουρα θα είναι σημαντικό σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει θρησκευτικών αξιών. Αυτό ωστόσο τώρα δεν έχει τεθεί ως ζήτημα, γιατί θεωρούμε ότι περιοριζόμαστε στο θέματα αστικού δικαίου και εμπορικού δικαίου. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε για θέματα οικογενειακού δικαίου. Αλλά ως τώρα δεν έχει τεθεί καν το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα, για το θέμα του θρησκευτικού δικαίου. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι γενικώ πώς αυτές οι αποφάσεις, με βάση αυτή τη σύμβαση, όπως και με βάση την εσωτερική ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, καταρχήν δεν ελέγχουμε τους κανόνες που εφάρμοσε η τρίτη χώρα. Η μόνη επιφύλαξη είναι η διεθνής ε, δημόσια τάξη. Ε, δηλαδή, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι τόσο συγκλονιστικό, ας πούμε, που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την απόφαση. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα σοκ που ε, αισθανόμαστε, γι' αυτό δεν εφαρμόζουμε την απόφαση. Ε, αυτό ισχύει σε όλα τα ε, δίκαια των κρατών μελών, ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με βάση αυτή τη Διεθνή Σύμβαση. Τώρα, τα στην περίπτωση του Ισλάμ, ας πούμε, ε, έχουμε το γαλλικό, ας πούμε, ακυρωτικό δικαστήριο. Ε, η πιο μεγάλη ε, μουσουλμανική κοινότητα, ας πούμε, είναι στη Γαλλία. το ακυρωτικό δικαστήριο μιλάει για το οικογενειακό δίκαιο, για την πολυγαμία, ας πούμε. αν η πολυγαμία έχει οικονομική επίπτωση, Φερρυπίν, αν δύο γυναίκες, ας πούμε, θέλουν ας πούμε, να μοιραστούν ε, ε, μία πολυκατοικία ας πούμε, ε, στη Γαλλία, εφαρμόζουμε την πολυγαμία ας πούμε, και το μοιράζονται. ενώ οι αποφάσεις ας πούμε, στο Μαγκρέμπ αντίστοιχε δεν αναγνωρίζονται. Εν πάση περιπτώσει, το σοκ μπορεί να μας οδηγήσει ή μάλλον το σοκ αυτό δεν ισχύει ποτέ για τα εμπορικά θέματα, εμπορικά αστικά θέματα. δεν θα υπάρξει αυτό το θέμα. Το βασικό θέμα που τίθεται στην πράξη είναι το θέμα της διαφθοράς ε, σε πολλές από αυτές ε, τις χώρες, ε, στο δικαστικό σώμα κτλ. Το θέμα είναι αν οι, οι λόγοι άρνησης αυτή τη στιγμή επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε αυτή τη δυσκολία που είναι συχνά κρυμμένη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα σε μια ε, απόφαση που έχει εκδώσει ένας διεφθαρμένος δικαστής από μια απόφαση που έχει εκδώσει ένας τίμιος δικαστής. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για, λιγάκι για το θέμα της Δανίας. Ξέρετε ότι η Δανία δεν συμμετέχει στην υιοθέτηση των μέτρων που ε, αφορούν την ε, αστική δικαστική συνεργασία. Δηλαδή, όταν υιοθετηθεί η σύμβαση τελικά και η Ένωση αποφασίσει να την ε, κυρώσει θα το κάνει η Ένωση, αλλά η Δανία θα το κάνει ως χωριστό συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση. Έχουμε μια παράλληλη συμφωνία όμως μεταξύ Δανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 και εκεί έχουμε κάποιες γενικές αρχές για τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και της Δανίας ε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις που επηρεάζουν τον κανονισμό Βρυξέλλες 1. Υπάρχει καλή συνεργασία με τη Δανία Για, να προσθέσω κάτι για την ερμηνεία αυτών των διατάξεων στη σύμβαση. Όπως ακούσατε τα, όσα είπε η Ανδρέα, ε, υπάρχουν και ειδικέ επιτροπές της σύμβασης που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και όπου όλα τα συμβαλόμενα μέρη συνέρχονται για να συζητήσουν θέματα ερμηνείας, την πρακτική εφαρμογή τη σύμβαση. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για να κατανοούμε ε, μονοσήμαντα τι διατάξει τη ε, ε σύμβαση για τι αποφάσει. Για τι ομαδικέ προσφυγέ. Δεν έχουμε ειδικού κανόνε. Αλλά η αρχή είναι ότι αν η απόφαση ε, σέβεται το δικαιοδοτικό φίλτρο, τότε ισχύει η σύμβαση και θα πρέπει να κυκλοφορήσει η απόφαση καταρχήν. Sí. Να διευκρινίσω μία πτυχή όσον αφορά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σχέδιο σύμβασης και τη διαιτησία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πράγματι εξαιρείται η διαιτησία γιατί υπάρχει και σύμβαση της Νέας Υόρκης που προβλέπει αναγνώριση και εκτέλεση. Αν πετύχαινε η σύμβαση. Ένας από τους στόχους, για παράδειγμα, της σύμβασης είναι οι δικαστικές αποφάσεις να μπορεί να διαθέτει και έναν παράλληλο μηχανισμό για να διασφαλίζει διασυνοριακά τις διάφορες δικαστικές ε, υποφάσεις. Οπότε μπορεί τελικά η δικαιοδοτική οδός να ευνοηθεί από τη σύμβαση αυτή. Και για τη δημόσια τάξη, ναι, φυσικά και περί αυτού πρόκειται. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με τη θρησκεία, στα εμπορικά ζητήματα παίζουν ελάχιστο ρόλο. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως το θέμα τη δημόσιας τάξη μπορεί να ενδιαφέρει, γιατί είναι θέμα αρμοδιότητας, ώστε να μην αναγνωρίζει αποφάσεις που να αντιβαίνουν στην αρμοδιότητα της. Υπάρχει και το άρθρο 10 της σύμβασης, το οποίο λέει ότι οι αποφάσεις που είναι τιμωρητικές και δεν πρόκειται μόνο για αποζημίωση, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στη δημόσια τάξη. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προδιαγραφές είναι τέτοιες που δεν θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τέτοιες τιμωρητικές αποφάσεις η κυρία Ζω. Ευχαριστώ. Πολλοί απάντησαν, αλλά έχω και εγώ να προσθέσω πράγματα για τις κοινέ προδιαγραφές και αρχές. Το σημείο εκκίνησης για την διατύπωση τέτοιων συμβάσεων είναι να βασίζονται σε κοινά αποδεκτές αρχές για να εφαρμόζεται όσο γίνεται ευρύτερα η σύμβαση. Οπότε γίνονται κοινά αποδεκτά κάποια πράγματα στην αρχή και πάνω εκεί χτίζουμε. Τώρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή. Υπάρχει το άρθρο 22 και 23 που λένε ότι η ερμηνεία πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Υπό την σύμβαση. Άρα η διεθνής ερμηνεία υπερέχει της εθνικής και η γραμματεία της Σύμβασης της Χάγης έχει επαφές με τις χώρες μέλη, οπότε συλλέγει δικαστικές αποφάσεις, νομολογία και έτσι η διάσκεψη της Χάγης και η γραμματεία συζητούν με την Ειδική Επιτροπή. τα συμβαλόμενα κράτη, ή ακόμα και αν δεν είναι ακόμα, κάθε 4-5 χρόνια ή και πιο συχνά αν χρειάζεται, συμβρίσκονται για να συζητήσουν τη λειτουργία της σύμβασης, πώς έχει πάει δηλαδή μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, ποια ήταν τα προβλήματα κλπ. Έτσι νομίζω ότι δημιουργούνται και οι κατάλληλες ερμηνείες. Τώρα, Έχουμε το αναφερουμένο κείμενο για την Ειδική Επιτροπή. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι δεσμευτικά, αλλά αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Άρα ο κόσμος θα καταλαβαίνει λίγο πολύ τι σημαίνουν οι διάφοροι όροι και θα μπορεί να έχει έτσι απαντήσεις. Για τις συλλογικές αγωγές όντως δεν αποκλείονται. Η εκτέλεση δεν αναγνωρίζεται βάσει τη σύμβαση. Οι αποφάσεις τώρα που έχουν πολιτική χρειά προβλέπονται και γι' αυτό και το άρθρο 7 δίνει τη δυνατότητα εξαιρέσεων και άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης. Σε θέματα όμως αστικά και εμπορικά μπορεί κάποιος να σκεφτεί το θέμα διαφωνιών ο κράτους επενδυτών. Τέτοιου είδους δικαστικές αποφάσεις έχουν πολιτική επιρροή και γι' αυτό δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της σύμβασης. Στα πλαίσια της διάσκεψης της Χάγης δεν προβλέπονται κυρώσεις για τις χώρες που δεν ακολουθούν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή δεν εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις που θα έπρεπε να εκτελέσουν. Αλλά υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία κάθε τόσο συνεδριάζει για να εκτιμήσει την κατάσταση. Και σε αυτά τα πλαίσια συζητούνται αυτές οι περιπτώσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Λεμπρετό για τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αιτιολόγηση άρνησης, πώς σταματάμε δηλαδή τις αποφάσεις ξένων χωρών να αποτελούν μέρος του εξοπλισμού των δικαστικών μας αποφάσεων. Έτσι όπως έχει συνταχθεί το άρθρο 7 αυτή τη στιγμή που εμπνέεται από την Σύμβαση του 2005 και έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί δηλαδή ευρωπαϊκό κεκτημένο, θέτει σωστά αυτή την ισορροπία, γιατί μπορεί να αποτρέψει δικαστικές αποφάσεις τρίτων χωρών να εκτελεστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως, προωθείται η εκτέλεση των ευρωπαϊκών δικαστικών αποφάσεων στο εξωτερικό. Εξαρτάται από τις περιπτώσεις, αν είναι θέματα δικαιοσύνης, την απόφαση δηλαδή, μερικές φορές τα δικαστήρια καλούνται να την εξετάσουν βάσει των συγκεκριμένων περιπτώσεων και όχι να την εφαρμόσουν ε, τυφλά. Ο κύριο Φω θέλει να ρωτήσει και κάτι ακόμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Όντω μια ερώτηση έχω να κάνω σε ό,τι αφορά τα δύο αυτά σημεία. Καταρχάς, Όντω. πώς ε, αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές αποφάσεις και έχω υπόψη μου για παράδειγμα την αντιπολίτευση στην ε, Ρωσία, την Τουρκία, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα κράτη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη λήψη πολιτικών ουσιαστικά αποφάσεων και εδώ θα πρέπει να μπει κάποιο όριο, να μην υποστηρίξετε, να μην το υποστηρίζουμε αυτό και από δική μας πλευράς να μην υποστηρίζουμε αυτά τα οποία δεν θέλουμε. Και ανακύπτει και το ερώτημα του τι ρόλο παίζει η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο κράτος λήψης της απόφασης. Είναι εντελώς ε, άσχετα το τι ρόλο παίζει η δικαιοσύνη. Και να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αμφισβητεί την ε, ανεκρατησία του κράτους. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αποδεχτούμε αυτά. Πρόκειται για θεμελιώδεις αρχές. όπου ουσιαστικά τι θα γίνει, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχουμε δυνατότητα αντιδράσει με κυρώσει. Σε περίπτωση που ένα κράτο μέρο δεν τηρήσει τι αρχέ μα. Επιστείω λοιπόν την προσοχή σε αυτό. Αν δεν υπάρχουν ε, επικυρώσει ε, αρχικά, ουσιαστικά μετά εξαρτάμαστε στην καλή θέληση των ε, ατόμων αυτών των κρατών αυτών. Και βάσει των εμπειριών μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι θα αποτελούσε μεγάλη αμέλεια. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την αντίδρασή μας σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εντάξει, τι να γίνει. Ακόμα και αν δεν υπάρχει εξαρτησία τη δικαιοσύνη στη χώρα αυτή, θα αναγνωρίσουμε τη δικαστική απόφαση. Κάπου θα, μπει, θα πρέπει να μπει ένα όριο. Γιατί πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να υποκρινόμαστε ότι δεν υπάρχει καν το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε κανένα εθελοντή. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να δώσω καθοριστική απάντηση φυσικά, αλλά να σας πω ότι έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Με διπλωματική γλώσσα προφανώς. Και εδώ θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το ποιον θα αφήσουμε να μπει. Και υπάρχουν όντως κάποιες χώρες που θέλουν να δημορφωθεί σε δημερές επίπεδο η συμφωνία αυτή. Δεν ήταν αυτή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιο σύστημα υπάρχει, για παράδειγμα, της ε, παιδιών, γιατί είναι τόσο ευαίσθητο, για παράδειγμα, το θέμα αυτό, που όσες ε, χώρες δεν έχουν ε, συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον θα μπουν ή όχι. Αλλά αυτό τελικά οδηγεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο συνονθήλευμα τιμερών συμφωνιών. Για το, δημε... το δεύτερο ερώτημα. Τι γίνεται αν εγκαταλείψει κάποιος μετέπειτα χρονική στιγμή την διάσκεψη, τη συνθήκη. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα δημόσιας τάξης ε, για να μην αναγνωρίσουμε την απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να προβούμε σε οριζόντια πράξη και να αποκλείσουμε τελικά τη χώρα αυτή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Καταρχάς σας ευχαριστώ που μένετε σε αυτό το στοιχείο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε τέτοια θέματα, προφανώς. Και δεν έχω να σας δώσω φυσικά οριστική απάντηση στο ερώτημα αυτό τώρα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το άρθρο 7 της, ε, του σχεδίου σύμβασης, όπως έχει ε, και μιλάει για τους λόγους άρνησης, ε, προβλέπει εντός του πλαισίου της σύμβασης κάποια εργαλεία που θα επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά εργαλεία να, την ανα... να αρνηθούν την αναγνώριση και εκτέλεση σε περίπτωση όπως αυτές που περιγράφεται, που είναι προφανώς σοβαρές περιπτώσεις. Μπορεί να μιλήσουν για δημόσια τάξη που δεν αφορμώ την εθνική δημόσια τάξη, αλλά και την ευρωπαϊκή. Διάφορα βασικά θέματα για μας, πολύ σημαντικά, όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή το γεγονός ότι η, απά, η απόφαση ε, προέκυψε μετά από μη δίκαιη δίκη ή μετά από απάτη. Και επομένως δεν ευθυγραμμίζεται με βάση τους δικούς μας δικαιοδοτικούς κανόνες ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα προβλέπει η σύμβαση. Και νομίζω ότι αυτέ οι περιπτώσει που είναι πραγματικά σοβαρέ, όπω αυτέ που περιγράψατε, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εντό του πλαισίου τη σύμβαση, χωρί να χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εκφύγει ε, του πεδίου τη ε, σύμβαση. Διαπραγματευόμαστε με την ιδέα ότι εμεί δεσμευόμαστε από αυτέ τι διεθνεί υποχρεώσει, δημιουργούμε ένα πλαίσιο όπου οι αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοστούν και σε τρίτες χώρες, αλλά και εμείς έχουμε τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε τα δικά μας δικαστήρια να προστατεύουν την, το ένομο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο λόγοι για αυτό το θέμα. Ε, από, την πλευρά, τη σκοπιά των ε, δικηγόρων. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης, πριν αναγνωρίσουμε μια ξένη απόφαση, φυσικά θα έχουμε μια ε, διαδικασία εκτελεστότητας. Σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτή τη διαδικασία, οι διάδικοι θα μπορούσαν εκ νέου να μιλήσουν όχι για την ουσία της υπόθεσης, αλλά να μιλήσουν για την πιθανή άρνηση εκτέλεσης. Μπορώ να σας πω ότι οι δικηγόροι θα προσέξουν πάρα πολύ το σεβασμό όχι μόνο της δημόσιας τάξης, του κράτους προς όνει αίτηση, αλλά όπως αναφέρει και η σύμβαση, στην περίπτωση που η διαδικασία που εφαρμόστηκε για να φτάσουμε στην απόφαση ήταν ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αρχές της δίκαιης δίκης και των δίκαιων ε, δικονομικών κανόνων. Περιλαμβάνεται η δημόσια τάξη αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Και βεβαίως η ανεξαρτησία της, ε, του δικαστικού σώματος και της δικαιοσύνης, ε, το κράτος δικαίου κτλ. Όλα αυτά είναι τμήμα. Αλλά συμφωνώ με τις ε, επιφυλάξεις ε, του καθηγητή Φιλιμπέρτη για την ε, διαφθορά κτλ των δικαστών. Υπάρχουν πράγματα που είναι κρυμμένα και δεν τα καταλαβαίνουμε με βάση την απόφαση έτσι όπως είναι γραμμένη και αποστέλλεται ας πούμε στο δικαστήριο του συμβαλόμενου μέρους, του συμβαλόμενου κράτους δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί για την εκτελεστότητα ή όχι. Πολύ γρήγορα Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία. Ε, άλλο πράγμα η διαφορά, έτσι. Η ανεξαρτησία. Κάποια μέρη, ας πούμε στην Τουρκία, στη Ρωσία, ε, όταν κάποιος είναι πολύ κοντά στην εξουσία, μπορεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Αλλά άλλοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Κάποιες εμπορικέ διαφορές δεν ε, επηρεάζονται καθόλου από την πολιτική κατάσταση. Ενώ άλλα δικαστήρια μπορεί να επηρεάζονται, να τα επηρεάζει ας πούμε, το καθεστώς. Μπορεί ας πούμε, να εκδίδονται αποφάσεις αυτές τις χώρες που δεν έχουν πρόβλημα ανεξαρτησίας των δικαστών. Έτσι, οι δικαστές εκδίδουν την απόφαση μια χαρά με βάση τις ανενόχλητη κτλ. Και για τα εμπορικά θέματα, η βασική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για να αποφύγουμε μια δικαιοδοσία που τη φοβόμαστε γιατί δεν υπάρχει ανεξαρτησία ή γιατί υπάρχει πιθανή δικαιος, ε, ε, διαφθορά είναι η προσφυγή στη διαιτησία. Έτσι λύναμε στο παρελθόν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό λοιπόν η διαιτησία για εμπορικά διεθνή θέματα έχει τόση επιτυχία γιατί αποφεύγουμε δικαστήρια όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση μικρή ή μεγάλη να υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες ας πούμε σε αυτά τα δικαστήρια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα. Δηλαδή δυνατότητα προσφυγή στη διαιτησία. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαντλήσαμε όλες τις ερωτήσεις, ακούσαμε και τις απαντήσεις. Εξαντλήσαμε και το χρόνο που προβλέπαμε για την ακρόαση αυτή. Οπότε ευχαριστώ πολύ τους ε, προσκεκλισμένους μας τους εξέχοντες προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με τα επόμενα σημεία. Dear Περνάμε στο σημείο 12 της σημερινής μας ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων έναντι τρίτων. Εγώ είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα. Οπότε επιτρέψτε μου να αρχίσω λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια που καλύπτει μια γραμμή που έχει να κάνει με το εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα χωρίσεων απαιτήσεων τετρίτων. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Ακόμα και αν το πεδίο εφαρμογής φαίνεται πολύ περιορισμένο, Οι εκχωρήσει απαιτήσεων έναντι τρίτων είναι κάτι που βρίσκουμε συνέχεια. Οπότε, ό,τι κάνουμε για αυτή την υπόθεση πρέπει να φροντίσουμε να το κάνουμε καλά. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο θέματα σήμερα. Το ένα είναι διαδικαστικό και θα πρότεινα να περιορίσουμε το έργο μας σε ορισμένα τμήματα μόνο της πρότασης της Επιτροπής. Το άλλο έχει να κάνει με την ουσία. Ποιες θα έπρεπε να ήταν οι επιλογές του εφαρμοστέου δίκαιου στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνει 15 άρθρα. Έχει να κάνει με τους κανονισμούς 1 και 2. Από ό,τι βλέπω εγώ, τα άρθρα 3 και 7 με 13 έχουν ληφθεί υπόψη χωρίς αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν θα επικεντρωθώ στα άρθρα 1 και 2, 4 με 6 και ίσως και στα τελευταία της πρότασης και σας παρακαλώ να κάνετε και εσείς το ίδιο. Το άρθρο 4, παράγραφος 1 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει τους κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για την κατοικία, τη συνήθη κατοικία. Τα νομικά συστήματα των χωρών μελών κανονικά δεν συμφωνούν για το ποιο πρέπει να είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Σε κάποιες χώρες μέλη το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της χώρας από όπου προέρχεται η αγωγή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι χώρες απέτησης, σε άλλες φορές εκεί που έχει γίνει σύμβαση. Οπότε θα έπρεπε να δούμε ποια τρίτα μέρη προστατεύουν αυτοί οι κανόνες. Τα τρίτα μέρη είναι οι πιστωτές συνήθως. Για τους πιστωτές η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η κατοικία προσφέρει περισσότερη διαφάνεια για τα τρίτα μέρη από την εναλλακτική του εφαρμοστέου δικαίου που έχει να κάνει με την ίδια την αγωγή. Εγώ λοιπόν θα συμφωνούσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κύριο κανόνα όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο σε τρίτους. Σε σχέση τώρα με απαιτήσει άλλες, η Επιτροπή προτείνει έναν ανορθόδοξο κανόνα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 που επιτρέπει τις δύο πλευρές σε συμφωνία να αποφασίσουν για το ποιο θα είναι το δίκαιο που θα εφαρμόζεται. Αυτό όμως αντιβαίνει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό το φως μάλιστα του άρθρου 3 θα ήταν σαν να πηγαίνουμε υπερβολικά μακριά. Πάντως η ρύθμιση θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε οι πλευρές που έχουν συμφωνήσει μπορούν να εφαρμόσουν το δίκαιο το οποίο έχει να κάνει με τις περισσότερες περιπτώσεις απαιτήσεων. Αυτά. Το θέμα είναι, έχετε σχόλια? Όχι από ό,τι βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο. Όχι, όχι. Ωραία. Οπότε τελείωσε αυτό το θέμα και συνεχίζουμε με το σημείο 13. Ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την τυχάσευση της παγκοσμιοποίησης, εμπορικές πτυχές. Εδώ η συγκεκριτής είναι ο κύριος Λεμπρετό. Κύριε Λεμπρετό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνεχάρη τον καθηγητή Κουνεπέρτη και τι μου υπενθύμησε ότι ήμουν καθηγητής του στην Γκρενόμπλ. Πολύ περήφανος είμαι λοιπόν, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι εγώ του έμαθα αυτά που ήρθε και μας είπε. Όντως, μας χαροποιεί αυτό. Ορίστε, το πρωί είδα κάτι συναδέρφους, τώρα συναντάω στις συνεδριάσεις με τους μαθητές μου ανησυχητικό αυτό, σημαίνει ότι γυρνάμε. Τέλος πάντων, έχω γνωμοδότηση για έκθεση της Επιτροπής ΙΝΤΑ όσον αφορά τον έλεγχο, τη διθάσευση της παγκοσμιοποίησης. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βασιζόμαστε σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο ετοίμασε στις 10 Μαΐου του 1917 που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Ενδιαφέρον γιατί η παγκοσμιοποίηση φυσικά και έχει πολλές θετικές πτυχές. Το υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εγγραφό της. Για παράδειγμα, κάθε δισεκατομμύριο εξαγωγών σημαίνει 14.000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάτι άλλο εντυπωσιακό. 30 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, δηλαδή η μία στις 7, εξαρτάται από τις εξαγωγές μας στο υπόλοιπο του κόσμου. Αυτό μας δίνει μια ιδέα για τη σημασία που έχει το ζήτημα. Και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι στο παραδοσιακό εμπόριο προσθέτουμε και το ψηφιακό εμπόριο όλο και περισσότερο, το οποίο μας υπόσχεται μεγάλο μέλλον. Όμως η παγκοσμιοποίηση έχει και κάποιες αρνητικές πτυχές. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθούμε σε dumping φορολογικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, υγειονομικό και μάλιστα κάποιες χώρες όπως η Κίνα μπαίνουν πολύ συχνά στο κάντρο αυτών των επιδεινώσεων σε διάφορους τιμής. Οπότε οι διεθνείς διαμάχες πώς θα επιλύονται. Τι δικαιοσύνη θέλουμε για να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του διεθνούς εμπορίου. Κυρίως διαφορές που φέρουν σε αντιπαράθεση τα κράτη με τους επενδυτές. Μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, δυστυχώ για να έχουμε απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα, έχουμε στη διάθεσή μας μία μόνο βάση. Έτσι ήθιστε. Και εγώ σκέφτηκα να επικεντρωθούμε σε τέσσερα σημεία για να αρχίσει η συζήτηση. Πρώτον, να λέμε ότι η παγκοσμιοποίηση πρέπει να σέβεται τις ευρωπαϊκές παραδόσεις. Κυρίως τις προστατευμένες την προστατευμένη προέλευση των προϊόντων. Πολύ βασικό αυτό και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Έχω την αίσθηση, είναι θέμα επικαιρότητα. Γιατί οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν σέβονται τέτοια ζητήματα. Θα θυμόμαστε για το TTIP, δεν ξεκινήσαμε καλά, όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον, μαζί σας μάλιστα πρόεδρε, είχα ρωτήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτέ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν χρειαζόμαστε καθόλου τέτοια ε, προστατευμένη ονομασία προέλευση. Ενώ η Γαλλία, τι, είναι μια χώρα μου δώσα να καταλάβω παλιωμοδίτικη. Εγώ δεν έχω καθόλου όμω αυτή την αίσθηση. Ενώ το ΣΕΤΑ, η συμφωνία μα με τον Καναδά, λαμβάνει περισσότερο υπόψη τι ονομασίε προέλευση και προστατεύονται από την συμφωνία αυτή. Τώρα, η μελλοντική συμφωνία με το Μεξικό που προετοιμάζεται αυτή την εποχή, από ό,τι έχω καταλάβει, η συμφωνία αυτή θα σεβαστεί ακόμα περισσότερο τις ονομασίες προέλευσης. Άρα η ανησυχία μας αυτή λαμβάνεται όλο και περισσότερο υπόψη. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, πρέπει να προστατεύσουμε την δημιουργία. Πολύ σημαντικό. Ο κύριο Καβαντά σήμερα το πρωί, σχεδόν ποετικά, αναφέρθηκε στο πλούτο της Ευρώπης που είναι ακριβώς η ικανότητα δημιουργίας. Συνεπώς πρέπει να προστατεύσουμε τη δικιά μας διανοητική ιδιοκτησία, τα δικά μας διπλώματα βρεσιτεχνίας. Τρίτο, σεβασμός δικαίου. Όταν το διεθνές εμπόριο που έχει βέβαια κανόνες, διαπιστώνουμε ότι παραβιάζονται αυτοί οι κανόνες, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στους δικαστές και έχουμε τρεις δυνατότητες. Μία όμως αναδύεται. Εθνική δικαιοσύνη, εγώ προσωπικά θα το προτιμούσα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Συχνά δεν εμπιστεύονται την εθνική δικαιοσύνη επενδυτές. Δεύτερον, τα διαιτητικά δικαστήρια. Τα τελευταία χρόνια αυτό προτιμήθηκε, αλλά έχουν χάσει την αξιοπιστία τους τελευταία. Γιατί αυτοί που αναλαμβάνουν τη διατησία συχνά έρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά δεν είναι αμερόληπτη και δεν έχουν διαφάνεια. Και η τρίτη λύση που επιβάλλεται είναι αυτή που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο προβληματισμού της, είναι ένα πολυμερές δικαστήριο επενδύσεων. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Σίγουρα καθυσυχάζει τους πάντες και τις χώρες και τους επενδυτές, γιατί οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και η διαδικασία διέπεται από περισσότερη διαφάνεια. Και το τέταρτο που ζητάω είναι να σεβόμαστε τις χώρες και τις αρμοδιότητές τους. Κύριε Ντίνα, δεν έχω ξεχάσει τα βασικά μου μαθήματα. Ξέρω ότι δεν ανησυχούσατε. Συμφωνώ με την Επιτροπή. Λοιπόν, πρέπει να σεβόμαστε την αρμοδιότητα των χωρών μελών. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι ελεύθερων συναλλαγών συνήθως προβλέπουν επιμερισμένη αρμοδιότητα και όχι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμερισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μέλη. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις αρμοδιότητες των χωρών μελών που υπενθύμησε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2017 για τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Άρα βαδίζουμε σε σίγουρα εδάφη. Πρέπει να υπάρχει πλαισίωση στην παγκοσμιοποίηση λοιπόν, γιατί κανείς μας ε, δεν θέλει μία παγκοσμιοποίηση χωρίς κανόνες. Θέλουμε μία φρόνιμη παγκοσμιοποίηση που να εντάσσεται σε νομικά πλαίσια στην υπηρεσία των εθνών και των ατόμων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Ο κύριος Ντυρό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν ε, παίρνω το λόγο για να α, σας πολεμήσω, αλλά για μια διευκρίνηση στο θέμα των δικαστηριών. Των πολυμερών δικαστηριών σε ό,τι αφορά τους επενδυτές. Είναι πραγματικά απαραίτητο, πιστεύετε, να υπάρχουν αποκλειστικές ε, δικαιοδοσίες για τα θέματα επενδυτών. Είναι μια ερώτηση για την οποία θα ήθελα μια απάντηση. Θα ήθελα μια απάντηση από τους ε, νομικούς, ο κ. Φως. Η δική μου ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση κινείται. Έχουμε συζητήσει διάφορε περιστάσεις για το TPTP, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Το θέμα των επένδυτων των ε, σχέσεων με το κράτος και πώς μπορεί να συμπεριληφθεί καλύτερα το θέμα αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα διεθνές δικαστήριο για να ασχολείται με τέτοια θέματα, προκειμένου να υπάρχει και εμπιστοσύνη σε τέτοια δικαστηρία και για να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Αυτά ήταν λοιπόν οι ερωτήσει προς τον κύριο Λεμπρετών. Θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ. Ναι. Το ίδιο ερώτημα ουσιαστικά ετέθησε και από τους δύο συναδέλφους το θέμα της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις διεθνεί επενδύσεις. Εγώ επαναλαμβάνω από προσωπικής άποψης, ε, θα, θα το προτιμούσα να δρά η εθνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό γιατί αν ακολουθήσουμε τη λύση αυτή, πολύ απλά δεν θα έρθουν πολλοί επενδυτέ. Γιατί εμεί τα βλέπουμε τα πράγματα από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη, όπου τα πράγματα λίγο πολύ λειτουργούν. Εν πάση περιπτώσει, όχι σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργεί. Αλλά ξέρουμε ότι πολλά εθνικά δικαστικά συστήματα δεν λειτουργούν σωστά. Η λύση λοιπόν που είχε προταθεί ως τώρα ήταν τα διαιτητικά δικαστηρία, γιατί έχει προχωρήσει πολύ το θέμα της διτητικής ε, δικαιοσύνης. Σήμερα όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε επιφλεκτικοί έναντι των ατόμων αυτών που είναι τόσο κοντά στους επενδυτές. Και βρισκόμαστε στην εξή παράδοξη θέση, όπου θα πρέπει να προστατεύσουμε τα κράτη από του επενδυτέ πλέον. Είναι μάλλον καινούργιο φαινόμενο. Και θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάτι διαφορετικό. Το οποίο ενδεχομένω να χρειαστεί φαντασία. Ενδεχομένω ένα διεθνέ δικαστηρίο με αξιόπιτου δικαστέ και με, μια διαφανή, τρόπο λειτουργίας. για να υποστηριχθεί αυτή η ιδέα η οποία έχει γίνει όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από όλους τους ακα... ακαδημαϊκούς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή ζήτησε το λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας ε, για την γνωμοδότηση αυτή. Να επισημάνω και κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω να μην σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με δικαστικά συστήματα. Βλέπουμε λοιπόν ε, μεγαλύτερο αποδεστισμό από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ και θέλαμε να τονίσουμε ότι θέλουμε φυσικά να ωφελήσουμε τον κόσμο. Δεν είμαστε αφέλεις βέβαια. Θέλουμε ελάχιστα πρότυπα για κοινωνικά ζητήματα και περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε στην καταπολέμηση αυτά με τον εγγονισμό, τον dumping από την Κίνα, τις ψευτοπιδοτήσεις από την Κίνα, αλλά και επενδύσεις από βασικές τεχνολογίες οι οποίες είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια ή για την αμοιβαιότητα. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας στην ανακοίνωση αυτή είναι ότι η παγκοσμιοποίηση μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν πρόκειται να εκλείψει. Χρειαζόμαστε λοιπόν συμφωνίες για να προωθήσουμε τις αξίες μας. Τις αξίες που μας καθιστούν ξεχωριστούς στην Ευρώπη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και τέλος, κάναμε άλλο ένα βήμα στην ε, διαφάνεια το TTIP παρά το γεγονό ότι αντιμετώπισε μεγάλη κριτική. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αυξήσει δραματικά την διαφάνεια. Είμαστε με μεγάλη διαφορά η περιοχή με τη μεγαλύτερη διαφάνεια στι συμβάσει τη. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποια σύσταση, έκανε τι συστάσει τη για την εντολή και θέλαμε και να κοινοποιήσουμε του λόγου ε, για την διαπραγμάτευση αυτή προκειμένου να τοποθετηθούν και εμπλεκόμενοι φορείς και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ γιατί φτιάξατε και το ευαίσθητο θέμα. του ότι α, μιας και οι επενδύσεις είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής, τίθεται το θέμα της προστασίας των στρατηγικών υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των επενδύσεων σε ε, υποδομές. Το θέμα λοιπόν αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, της εμπορικής πολιτικής και νομίζω ότι στο σημείο αυτό εξαρτήσαμε και το θέμα αυτό και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών. Άρα όλοι όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν στο θέμα αυτό, παρακαλώ να φύγουν από την αίθουσα.